να αυτά τα δύο να τα δούμε μαζί. Είναι σημεία που είναι συνδεμένα μεταξύ τους, έχουν σχέση. Έτσι, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, αυτό και θα κάνουμε. Το σημείο 2, τα έγκριση των πρακτικών τη 1 η και 2 Δεκεμβρίου του 2009. Θα εγκριθούν στο τέλος ε, της συνεδρίας αυτής, από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει κάποια παρατήρηση από δική σας πλευράς. Το σημείο 3 να σας πούμε ότι οι συντονιστές συναντήθηκαν και στην τελευταία τους συνάντηση εξέτασαν την ανακοίνωση της Επιτροπής ε, για τη θέση της ισχύ, σε ισχύ της συνθήκη της Αβώνας ε, και για τις διαθεσμικές ε, μεταβολές που τη λήψη αποφάσεων και θα πρέπει να εγκριθεί και η πρόταση, πρέπει να εγκριθούν οι προτάσεις εκτός από το συνταξιοπατήριο δικαίωμα και τη μεταφορά του. Κύριε Βανχόιτεν ε, θα πρέπει να μας ενημερώσει, δεν είναι όμως μαζί μας και θα συναντηθούμε μαζί της, θα δούμε για την ενδεχόμενη μεταβολή νομικής βάσης, μάλλον από τη στιγμή που υπήρξε αλλαγή της νομικής βάσης, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και τη θέση μας ε, και να έχουμε μια νέα τοποθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου Είναι η οδηγία για τον ε, χρόνο εργασία και κανονικά είχε ε, λήξει αυτό το θέμα και δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Κάτι ακόμα που θα πρέπει να σα προτείνω είναι να φτάσουμε στο κεντρικό πυρήνα της εργασίας μας που είναι το σημείο 4 και τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων εγγύων, λεχόνων και γαλουχουσών γυναικών η κυρία Ρόβανα Πλάμπ, η συγγήτρια, έχει το λόγο για να δούμε και τις τροπολογίες. Αύριο θα ψηφίσουμε. Πριν λάβει το λόγο λοιπόν θα ήθελα να ευχηθώ το καλό ορίσατε στον κύριο Τσούπα Τσαντόρ που είναι στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο στο Φιντές βουλευτής και υπεύθυνο σε θέματα παρόμοια στο Κοινοβούλιο Έχετε το λόγο κυρία μου.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 θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον που έδειξαν σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Τόσο σημαντικό για τις γυναίκες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη βελτίωση των ε, συνθήκων εργασίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, τα προβλήματα αυτών των γυναικών και να μπορέσουμε να αποκατέσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και στην οικογενειακή και αυτό για να βοηθούμε και στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να σας πω κάτι. να σας πω ότι οι πολιτικές ομάδες ε, πέτυχαν μια συμφωνία για την περίοδο αυτή άδεια μητέρων ε, και για τα επιδόματα σχετικά με αυτή την άδεια, επίσης και για τις υπόλοιπες συνθήκες οι οποίες ισχύουν ε, που έχουν να κάνουν αποκριστικά με την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία των γυναικών αυτών και να εγγυηθούμε την προστοθία όλων των εργαζομένων γυναικών, εγγύων, λεχώνων και γαλουχουσών. Για τη διάρκεια της Μητρικής άδεια η πρόταση της δικής μας ομάδας ήταν ε, να ισχύει για 20 τώρα μήνες αντί για 18 που ισχύει πριν που ισχύει πάντα μάλλον και όπως προτείνει η Επιτροπή και ακόμη για τα επιδόματα κατά τη διάρκεια αυτής της μετρικής άδειας εμείς προτείναμε ένα full payment όπως το αποκαλούμε για αυτήν την ε, διάρκεια της μετρικής άδεια και έτσι η διαφορά ε, πληρωμής ε, αποζημίωσης ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες να μην υπάρχει και να μην τιμωρούνται μέσα οι γυναίκες μόνο και μόνο επειδή γεννούν. Τώρα για την ε, πατρική άδεια. Εδώ είχαμε μία μεταβολή στην, ε, στο σκεπτικό 13 της πρότασης της Επιτροπής και εκεί αναφέρεται ότι επίσης και οι πατέρες έχουν δικαίωμα ε, να κάνουν χρήση μιας πατρικής άδεια ακριβώς. Και εμείς αυτό που προτείναμε είναι μία, προ, μία περίοδος έξι εβδομάδων μετά τον τοκετό και οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες ζήτησαν μια υποχρεωτική περίοδος άδειας πριν από τον τοκετό τεσσάρων εβδομάδων ή δύο εβδομάδες πριν ακριβώ τον τοκετό. και μετά από την ε, προσπάθεια για την επίτευξη συμβαστικής λύσης ε, και την ε, κατάλληλη ψηφορία που δόθηκε πριν από τις δύο ώρες στους αδέλφους, εμείς συμφωνήσαμε σε αυτή τη συμβαστική λύση και περιμένουμε πάντα μία απάντηση σε ένα θέμα και μόνο που έχει να κάνει με με, τους έξι μήνες υποχρεωτικής ε, άδεια ε, και που θα εφαρμοστεί για τις εργαζόμενες ε, γυναίκες ε, ασχέτως των ημερών άδεια πριν από το τοκετό και περιμένω επ' αυτού τη σύμφωνη γνώμη άλλων πολιτικών ομάδων. Περιμένω επίσης τις απαντήσεις λοιπόν των πολιτικών ομάδων στα πλαίσια της Επιτροπής μας έτσι ώστε να δω τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Εδώ θεωρώ ότι η περίοδος 18 εβδομάδων για τη μητρική άδεια και την πλήρη αποζημίωση που έχει να κάνει ακριβώς με αυτήν την περίοδο μητρικής άδειας νομίζω ότι αποτελούν πρόοδο η οποία επιτυχάνεται με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και τη δυνατότητα επιστροφής στην αγορά εργασίας επανόδου και την ε, δική εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασία, ε, ταυτόχρονα όμω με κείμενα και το δικαίωμα φύλαξη των παιδιών. Και εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι είμαστε και υπεύθυνοι απέναντι στου πολίτε, στου Ευρωπαίου. Θα πρέπει να θετήσουμε τα σημεία αυτά αυτές τις προτάσεις και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νομίζουμε ότι θα κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός υπέρ των πολιτών. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και Μέρ, ξεκινάει να σας πω, α, μισό λεπτό, στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας, ε, μάλλον ε, κοινή εταιρική. Θα πρέπει να συνηθίσουμε στην αερολογία. Ακούστε κύριε μου να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Γκρούνινγκ ε, Σκιώδη Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη για την καθυστέρησή μου, αλλά αντιμετωπίσαμε τρομερά προβλήματα για να ανέβουμε με τα σανσέρ και να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν περνούσαν, δεν μας έπαιρναν. Να σας πω όμως ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν προτεραιότητα για να μπορούν να έρθουν εδώ να μπαίνουν στα σανσέρ. Δεν έχω τα κείμενά μου. Γι' αυτό ό,τι θυμάμαι θα σας πω. Με την κύριε Πλάμβο και ε, εργαστήκαμε από κοινού, συνεργαστήκαμε και συμφωνήσαμε για την περίοδο 18 εβδομάδων με πλήρη καταβολή αυτού του, του επιδόματος ε, μητρότητας και για την περίοδο αυτής της ε, άδειας είμαστε σύμφωνοι για τις υποχρεωτικές έξι εβδομάδες ε, μετά τον τοκετό και τις δύο εβδομάδες ε, υποχρεωτική άδεια πριν από τον τοκετό. Δεν προτείνουμε την ψήφιση όλων αυτών των τροπολογιών που έχουν να κάνουν με την ε, πατρική άδεια, δεν είναι αυτό το οριστικό κείμενο, θα υπάρχει ένα άλλο κείμενο για τις γονικές άδειε και θα, έχει, θα ασχοληθεί και με την πατρική άδεια εκεί και για τις απολύσει κάτι υπέρ μιας τροπολογίας μάλλον είμαστε που θα προστάτευε την ε, νεαρή γυναίκα όταν επανέρχεται στην εργασία της ε, για δύο εβδομάδες ε, μετά την επάνωδό και έτσι ε, πριν, τρεις εβδομάδες πριν το ανακοινώνει αυτό στον εργοδότη της ε, και τον κύριο Τόμας Μαν την τροπολογία υποστηρίζουμε επίσης ε, που έχει να κάνει με τη συμπερίληψη των ανεξαρτήτων των ελεύθερων επαγγελματιών σε αυτό το κείμενο αλλά σε ένα άλλο κείμενο που θα ήταν καλύτερα προσαρμοσμένο. Αυτά θα ήθελα να σας πω για τα κύρια σημεία Βέβαια για το πρόβλημα κατάθλιψης κάπως ε, μετά από τον τοκετό, εντάξει συμφωνούμε, να μην συμπεριληφθεί αυτό στη μετρική άδεια και επίσης ε, δεν θα ε, υποστηρίξουμε την τροπολογία για την υποχρεωτική θύλαση παιδιών σε δύο χρόνια. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω σε όλο τον κόσμο εδώ που μας κάνει την τιμή να έρθει εδώ να παρακολουθεί τη συνεδρίασή μας και είναι όρθιο όμως η 1G3 εκεί αναμεταδίδεται ακριβώς η συνεδρίασή μας μπορούν να πάνε και να βρουν και θέση να καθίσουν εκεί. Λοιπόν, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι εάν κάποιος συνάδελφος σήξει το εξή θέμα. Εάν δηλαδή αυτό που συζητάμε είναι σωστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα, ένα που να μπορούν να το φορέσουν όλοι δηλαδή. Πιστεύω ότι αυτή η ρύθμιση δεν χρειάζεται, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχουμε ένα θαυμάσιο καθεστώς για την προστασία των εγγύων εργαζομένων γυναικών. Λειτουργεί θαυμάσια. Έχουμε επίσης ε, και εκπροσώπους στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο που έχουν ε, εργαστεί όντας έγκυες και δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε οτιδήποτε στην ε, νομοθεσία. Φαίνεται ότι σε ορισμένε χώρε το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, οπότε έγκυται στη διακριτική του ευχέρεια να εφαρμόσουν τους ε, κανονισμούς που χρειάζονται και το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται και δεν βλέπω γιατί θα πρέπει εμείς να ανακατευτούμε. Ε, και δι, το κόστος αυτό θα είναι πάρα πολύ υψηλό και θα επιβαρυνθούν οι εργοδότες δεν λέω ότι ορισμένοι εργαζόμενοι χρειάζονται συγκεκριμένα ωφέλη, αλλά θα πρέπει να είναι κοινωνικό το κόστος αυτό και όχι να το φορτώσουμε στις πλάτες συγκεκριμένων εργοδοτών για τους οποίους το βάρος αυτό θα είναι πάρα πολύ βαρύ. Ιδίω στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Κροκοδίλια δάκρυα χύνουμε για τα βάρη και τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά εδώ πρόκειται να ψηφίσουμε ένα πλαίσιο ρυθμιστικό το οποίο θα τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Και βεβαίως δεν λέω ότι δεν πρέπει να λάβουν μια ε, άδεια ε, μετά την ε, αφού αποκτήσουν το, το παιδί, αλλά ορισμένες ε, γυναίκες δεν ε, επιθυμούν να γυρίσουν στην εργασία. Είναι ε, λυπηρό επίσης, και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, δεν συμφωνώ, μεν, αλλά πολλοί εργοδότες δεν θέλουν να προσλάβουν νιόπαντρες ή γυναίκες έγκυες, διότι ξέρουν ότι ενδέχεται να μην επιστρέψουν στην εργασία τους. Εάν λοιπόν εμείς εδώ διακόπτει η πρόεδρος Μπορώ ναι. να σας διακόψω. Να σας διακόψω, γιατί εδώ δεν συζητάμε επί της ουσίας. Συζητούμε επί των τροπολογιών. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν έχετε σχολιάσει καθόλου τροπολογίες. Ή θα σχολιάσετε τροπολογίες ή δυστυχώς θα πρέπει να σας αφαιρέσω το λόγο. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ολοκλήρωσα τις παρατηρήσεις μου και ευχαριστώ για τα σχόλια που μόλις κάνατε. Κυρία Κορνέλισεν. Yeah, I was a bit surprised. Ναι, με εξέπληξε το γεγονός της διαδικασίας που ακολουθείται σε αυτή την γνωμοδότηση. Συνήθως ε, γίνονται ε, διαβουλεύσεις μεταξύ των σκιωδών εισηγητών σε γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις ε, μίζωνος σημασίας και δεν νομίζω να έχει γίνει αυτό μέχρι τώρα, τουλάχιστον δεν έχω ενημερωθεί. Μπορεί να έχουν γίνει διαβουλεύσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αν είχαν συμμετάσχει όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Άλλη μια παρατήρηση που αφορά τον κατάλογο ψηφοφοριών, ψηφοφορία, συγγνώμη, που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μπερδεμένος ε, ε, όσον αφορά την ε, σειρά των τροπολογιών αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει ο κατάλογος τροπολογιών, θα πρέπει να ψηφίσουμε εναντίον μια τροπολογία την οποία όμως υποστηρίζουμε εάν δεν περάσει μια άλλη τροπολογία που προηγείται. Ε, υπάρχει λοιπόν μια σύγχυση στον κατάλογο και πρέπει να τον αποσαφηνίσουμε. Αυτή η έκθεση είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντική και την έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Οι πράσινοι, η κυρία Στρέλα, την υποστηρίζουν πλήρως και θα ήταν κρίμα ε, αν αποδυναμώσουμε την ε, έκθεση ε, της Επιτροπής Γυναικών αντί να την υποστηρίξουμε. Γι' αυτό δεν θα μπορέσω να υποστηρίξω μια γνωμοδότηση η οποία ενδέχεται να αποδυναμώσει την έκθεση της Επιτροπής Γυναικών. Όσον αφορά την άδεια πατρότητας, υπάρχει μια ίση ε, διαίρεση, ίση κατανομή του βάρους μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει να έχουν και όλοι οι πατέρες, είτε ναι είτε όριμοι σε ηλικία, να έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον τις πρώτες ε, εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού τους να μάθουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, να είναι κοντά στο νέο γέννητο, να μάθουν να το πλένουν, να ασχολούνται και να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν την καθαριότητα, τη ρουτίνα του κλπ. Εάν θέλουμε στις κοινωνίες μας αυτές που γυράσκουν να ασχολούνται και οι δύο γονείς με τον νεογέννητο θα πρέπει να καταστήσουμε την περίοδο αυτή ελκυστική και να διαθέτουμε να δίνουμε ίσο βάρος και στην άδεια μητρότητας και στην άδεια πατρότητας. Εν συνεχεία, η προστασία κατά των διακρίσεων και κατά της ε, άδικης απόλυσης, αθέμητης ε, απόλυσης των εργαζομένων. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε τη δυνατότητα οργανισμών να αναλαμβάνουν την εισπεράσπιση περιπτώσεων όπου έχουν σημειωθεί διακρίσεις κατά εργαζομένων. Έχω συζητήσει με έναν διευθυντή μιας υπηρεσίας κατά των διακρίσεων και μου έχει εξηγήσει πώς της ζωτικής σημασίας είναι αυτή η αποφογή και καταπολέμηση των διακρίσεων. Παρακαλώ λοιπόν, μην το διαγράψετε, μην το αποδυναμώσετε και τέλος θα πρέπει οι άδειε μητρότητος και πατρότητος να πληρώνονται στο 100%, δηλαδή να λαμβάνουν το 100% της αμοιβή πληρωμής της αποζημίωσης. Ε, ανεξάρτητα από το εισοδηματικό του επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι μπορούν να, να έχουν ένα παιδί ή περισσότερα όπως το επιθυμούν. Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με τον κατάλογο ψηφοφορία, ελήφθησαν ήδη υπόψη τα σχόλιά σα και έχει ληφθεί η απαραίτητη μέρημνα. Δηλαδή, πρώτα θα ψηφιστούν οι τροπολογίε, ε, οι οποίε είναι συμβιβαστικέ τροπολογίε και μετά θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε, ξεκινώντα από τι τροπολογίε εκείνε που είναι πιο απομακρυσμένε από το κείμενο. Κυρία Ήρσπη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συνεργασία της, ιδίω σε αυτό το θέμα όπου είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε το θέμα από κοινού και να μην ε, μείνουμε αμετακίνητοι ε, σε παγιωμένες θέσεις πιστεύω ότι 18 εβδομάδες είναι μια σωστή προθεσμία, μια ισορροπημένη χρονική περίοδος η οποία ε, διαφυλάτει τα συμφέροντα και των εργοδοτών και των εργαζομένων. Όσον αφορά τώρα την ε, ε, οικονομική αποζημίωση. Εδώ αναφέρω ε, το, σύνθημα ίση πληρωμή, equal pay. Θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε αυτά. Επίσης, συμφωνούμε με την ε, άδεια μητρότητος μετά βεβαίως από την γένα, αλλά και πριν από την ε, ε, γέννα θα πρέπει η γυναίκα να έχει ένα ε, διάστημα χι εβδομάδων εκτός εργασίας. Αυτό δεν είναι καθιερωμένο σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν είναι ίδιο, ίδια η χρονική περίοδος αυτή. Πρόκειται εδώ για την προστασία της υγείας των εγγύων γυναικών και Γι' αυτό πιστεύουμε ότι διευρύνουμε το πλαίσιο αυτό προστασίας και διασφάλισης ε, των καλύτερων συνθήκων. Ε, θα απορρίψουμε μερικές τροπολογίες ε, οι οποίες αντιτίθενται στην εργασία αλλά συγχρόνως με τη δυνατότητα απόκτησης παιδιών και ανατροφής των παιδιών. Ε, τροπολογίες που έχουν αρνητική προσέγγιση θα τις απαρρίψουμε. Επίσης, είχαμε προτείνει και ορισμένες ε, τροποποιήσεις, ε, ορισμένες τροπολογίες όσον αφορά τις διάφορες εκστρατείες για τα θέματα της υγείας και το ενδεχόμενο της ε, κατάθλιψης ε, μετά από την ε, γέννηση του παιδιού, τη δυνατότητα δηλαδή να προσιαστεί αυτό το φαινόμενο. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες έτσι ώστε το βάρος της απόδειξης μπορεί, επειδή μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις κατά τα γυναίκα. πρέπει να το εξετάσουμε πιο σοβαρά. Ορισμένες τροπολογίες αφορούν πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Παραδείγματο χάρη όταν τα παιδιά δουν το φως της ημέρας με, με ορισμένες ε, εβδομάδες καθυστέρησης ή όταν γεννηθούν με ειδικέ ανάγκες εδώ θα πρέπει να εφαρμόσουμε ε, μεγαλύτερες ε, χρονικές περιόδους, δηλαδή να διευρύνουμε τις προθεσμίες αυτές, δεδομένου ότι υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις με ειδικές ανάγκες και να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη σε αυτές οι ε, συγκεκριμένες περιστάσεις. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε, μία, σε ένα συμβιβασμό. Αυτό που έχει σημασία είναι να δεχθούμε ε, τις τροπολογίες οι οποίες ε, είχαν μέχρι τώρα μία αρνητική προσέγγιση ορισμένα κράτη-μέλη και να πείσουμε το Συμβούλιο να ακολουθήσει τη γραμμή μας. Ο κύριος Τόμας Μάν. Η κυρία Φιγκερέδο όμως πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ε, έχω κάποιες αποσαφηνήσεις. Γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς προς ποια κατεύθυνση οδεύουν οι, τροπολογίες, ή, συγγνώμη, οι τροπολογίες. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν ε, μας έχουν κοινοποιηθεί ε, και είναι σημεία τα οποία βασίζονται στις 18 εβδομάδες. Θέλω να ξέρω λοιπόν τι έγινε και ε, θα ήθελα να μας εξηγήσει η συγγήτρια πώς έφτασε σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Διότι, διότι ε, ξέρετε, η γνωμοδότηση που θα ε, προκύψει εδώ θα δεν θα ακολουθεί την ίδια οδό με την έκθεση Εστρέγια. Και βεβαίως αυτό δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών είχε εκπονήσει και υιοθετήσει έκθεση βάσει των προτάσεων της ε, Edit Εστρέγια που ακριβώς ανέφερε τις 20 εβδομάδες ε, πληρωμένης άδειας μητρότητος. Όσον αφορά δε την άδεια ε, πατρότητος, ε, αυτή ανεφέρεται ως αναφέρετο δικαίωμα της γυναίκας να συνεχίσει να εργάζεται και ως επίσης εξίσου αναφέρετο δικαίωμα των πατέρων να ασχολούνται με τα παιδιά τους από τη στιγμή της γέννησής τους. Την δυνατότητα λοιπόν που θα έχουν οι μητέρες εάν το επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται και αντίστοιχα οι πατέρες να ασχολούνται με τα παιδιά τους. Η άδεια μητρότητος λοιπόν και η άδεια πατρότητος ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούν τις αναφορές εκθέσεως της Εντίτε τρέγια». 20 εβδομάδες λοιπόν, 20 εβδομάδες οι οποίες πρέπει να σας ομολογήσω ότι μου είναι ιδιαίτερος προσφυλής και επίσης θα ήθελα ιδιαίτερη μνήμα να γίνεται στην ε, περίπτωση γυναικών, εγγύων γυναικών που αντιμετωπίζουν ε, την απόλυση. Γιατί νομίζομαι ότι θα πρέπει πραγματικά να βελτιώσουμε την πρόταση οδηγίας ε, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια κατάσταση που θα είναι πραγματικά διαφορετική από την κατάσταση την οποία αντιμετώπιζε η οδηγία πριν από 17 ή 20 χρόνια. Ε, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι το ποσοστό ε, γεννητικότητας είναι πάρα πολύ χαμηλό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τώρα είναι η στιγμή να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε η μητρότητα και η πατρότητα να γίνει πιο ελκυστική και να αποτελέσει ένα θεμελιώδες κοινωνικού δικαίωμα του οποίου οφείλουμε να υπεραμεινθούμε. Δεν είναι δυνατόν τώρα να οπισθοδρομήσουμε. δεν είναι δυνατόν τώρα να πούμε καλά δεν πειράζει, καλή ήταν η κατάσταση και 16-17 χρόνια πριν, ε, ας μην προχωρήσουμε παραπέρα. Όχι, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να αποσαφινιστούν. Ευχαριστώ πολύ. Τόν μας Μάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα διαφοροποιηθώ από την ε, κυρία Φεραίρο. Εάν θέλουμε ε, να ενισχύσουμε την απόφαση μια άλλη επιτροπή, τότε δεν χρειάζεται η διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία. Α το αποφασίσει η άλλη επιτροπή και εμεί και θα γνωστοποιηθεί σε εμά. Εφόσον υπάρχει συνεργασία, ένα πλαίσιο συνεργασία, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές θέσεις. Κυρία Φιγκερέρο, ε, μην ξεχνάτε ε, ε, το σημείο εκκίνησης πριν, ε, πολύ πρόσφατα, ορισμένοι υποστήριζαν 14 εβδομάδες και ούτε μια μέρα παραπάνω. Άλλοι υποστήριζαν 21 εβδομάδες. Και η κυρία Γκρουνή ως ε, ε, συντονίστρια και από τους φιλελεύθερους επιτύχαμε έναν συμβιβασμό έναν, για να επιτύχουμε τον κοινό στόχο. Δεν ήταν καθόλου απλή αυτή η διαδικασία. Ήταν δύσκολη και χρονοβόρο, αλλά το επιτύχαμε και πιστεύω τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά. 18 και πλήρης ε, αμοιβή ε, πιστεύω μπορούμε όλοι να ζήσουμε, όλοι να το δεχτούμε. Ακούω πάλι τα ίδια παράπονα. Πατρική άδεια, πατρική άδεια. Βεβαίως μα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν μπορούμε όλα εδώ να τα συγκεράσουμε, όλα στο ίδιο, στο ίδιο καζάνι να τα ρίξουμε. Είναι τελείως λανθασμένη, λανθασμένη αυτή η προσέγγιση. Το θέμα της άδειας πατρότητος πρέπει να το εντάξουμε κάπου αλλού, σε ένα άλλο σημείο, σε μια άλλη γνωμοδότηση. Όχι όλα μαζί να τα ρίξουμε στο ίδιο σακί, διότι στο τέλος δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τίποτα και θα επικρατήσει μια χαόδης κατάσταση και θα, όλοι θα χάσουν. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα που συζητάμε εδώ. Κάποτε στο σχολείο <laughs> πήρα ένα πάρα πολύ καλό βαθμό γιατί είπα ότι το θέμα είναι άσχετο που μας δίνεται, αλλά εν συνεχεία εντάξει, τα φτιάξα με τον δάσκαλό μου. Λοιπόν, μην το κάνουμε αυτό. Α, τώρα, τι γίνεται ε, με το 101-102. Η κυρία Πλάμπ, ε, μιλήσαμε μαζί της και εγώ πιστεύω και το λέω στα αγγλικά ότι θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλη μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης αμοιβή. Άρα θα πρέπει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους πόρους για να μπορέσουν να καλύψουν αυτήν την διάταξη, αυτή την απέτηση. Έτσι λοιπόν μπορώ με τη διατύπωση αυτή μπορώ να συμφωνήσω. Επίσης δύο εβδομάδες πριν από τη γέννηση και έξι εβδομάδες μετά και αυτή είναι μια πρόταση, όπως το είπε και η κυρία ε, Γκρούνε, μπορούμε να δεχτούμε αυτή την πρόταση. Εάν διατηρήσουμε αυτή τη θέση σταθερή θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα γενικό συμβιβασμό και θα παρουσιάσουμε και μια πολύ καλή εικόνα της Επιτροπής μας ε, προς το κοινό, προς τη δημοσιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Euh, euh, euh, κύριε Κέτλερ και μετά κύριε Στρέλια. Ε, Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα μιλήσω από γερμανική σκοπιάς. Είμαι και πατέρας δύο παιδιών. Στη Γερμανία έχουμε ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί θαυμάσια. Πιστεύω ότι είναι στην κορυφή των κοινωνικών ε, παροχών του κοινωνικού πλαισίου στην Ευρώπη. 100% ε, αμείβονται όσοι, ε, οι λεχόνες ε, οι οποίες έχουν άδεια και πιστεύω ότι δικαιούνται απολύτως μια οικονομική, την οικονομική αποζημίωση διότι είναι και ο στόχος μας να πληρώνονται οι ε, γυναίκες αυτές, οι λεχόνες δηλαδή δεδομένου ότι είναι πολύτιμες γενικά για την εργασία και για την οικογένεια. Εάν εφαρμόσουμε εδώ το κριτήριο της... Ε, Sehr της επικουρικότητας, Πιστεύω ότι αυτή η λύση είναι πολύ ικανοποιητική και μπορούμε να δώσουμε τη διακριτική ευχέρεια στα εθνικά δίκαια, στις εθνικές νομοθεσίες, να ε, μεταβάλουν, διορθώσουν, βελτιώσουν και ενισχύσουν τις εθνικές τους θέσεις. Δεν μπορούμε όμως να δώσουμε ε, ε, ε, το έναυσμα στη δική μου χώρα, στη Γερμανία, να ξαναρχίσει φτούχια από την αρχή όλες αυτές τις συζητήσεις για τις διατάξεις οι οποίες αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της γερμανικής νομοθεσίας λειτουργούν ως πρότυπα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στις θέσεις αυτές που προτείνονται και να μην αλλάξουμε τίποτα. Κυρία Εστρέλια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θα ήθελα να σας πω το εξής, ε, να σας ε, πω για δύο-τρία στοιχεία που μου φαίνονται σημαντικά. Η οδηγία αυτή η οποία αναθεωρείται ε, βγήκε 17 χρόνια πριν και η νέα οδηγία θα διαρκέσει, θα ισχύσει για λίγο παραπάνω από μία δεκαετία. για το μέλλον εμείς νομοθετούμε και όχι για τώρα. Το δεύτερο στοιχείο, τι αφορά τις προκλήσεις τις δημογραφικές που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και την ανάγκη που αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη-μέλη, το γνωρίζει άλλωστε η Ευρώπη, να πρέπει να παροτρύνουν τον κόσμο τους για την αύξηση της γεννητικότητας. Αναγνωρίζουμε όλοι μας ότι θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό γεννητικότητας και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την συνθήκη της Αβώνας και την Ατζέντα 2020-2020 από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχουν διεξαχθεί έρευνες, όπως επίσης και από ανεξάρτητους οργανισμούς και το συμπέρασμα ήταν ότι για να βγει κανείς από την οικονομική, δημοσιονομική κρίση, στην οποία τώρα είμαστε βυθισμένοι, είναι πολύ σημαντική η παρουσία των γυναικών γι' αυτό για να λυθούν τα προβλήματα στην αγορά εργασίας για τις διάφορες χώρες ε, σίγουρα θα πρέπει να συνεισφέρουν και οι γυναίκες ε, για την οικονομική τους ανάπτυξη. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά να αναφέρω τρεις σημαντικές ε, αρχές. Πρώτα απ' όλα, μη διακρίσεις. Πρώτο σημείο σημαντικό η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών έχει σαν στόχο να προωθεί τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες και να δίνει μάχη κατά οποιασδήποτε διάκριση. Και εγώ είμαι συγγήτρια. Επίσης, δεν θέλουμε και διακρίσεις κατά των ανδρών και οι πατέρες θα πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα να συμμετέχουν στην στο μεγάλωμα των παιδιών τους, να μπορούν να παρακολουθήσουν ακριβώς τα παιδιά τους ε, στην πορεία τους ε, και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στην οικογενειακή ζωή και ο ρόλος των πατέρων λοιπόν. Και επίσης ε, και για τα παιδιά τα ίδια είναι πολύ σημαντικό να έχουν και τους δύο γονείς και τον πατέρα και τη μητέρα. Και κάτι ακόμα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να υπάρχει διάκριση στην αγορά εργασίας κατά της γυναίκας και να θεωρείται σαν μια εργαζόμενη δεύτερης κατηγορίας. Όχι μόνο γιατί κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες. Ξέρετε ότι το χάσμα, η διαφορά πληρωμής αμοιβή από άνδρα σε γυναίκα είναι περίπου στο 17% μέσος όρος. Αλλά ταυτόχρονα να μην ακούγονται αυτά τα στερεότυπα ότι οι γυναίκες ε, είναι δεύτερης κατηγορίες και μπορούμε και να μην τις υπολογίζουμε στην αγορά εργασία. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να περνάει έτσι εύκολα αυτή η ιδέα. Σχετικά με τις αμοιβέ. Θα πρέπει να πληρώνονται οι άδειε αυτές ε, στο 100% και ε, έτσι αυτό αποτελεί και μια παρότριση η αύξηση των γεννήσεων. Αν είχαμε μια μείωση του εισοδήματός τους επειδή γεννούν παιδιά, αυτό θα ήταν αρνητικότατα, γιατί ακριβώς ε, η γέννηση ενός παιδιού συνεπάγεται και αυξημένο κόστος, περισσότερα έξοδα για την οικογένεια. Κάτι ακόμα, να δούμε τη διάρκεια πριν από 17 χρόνια η διάρκεια της άδεια ήταν 14 εβδομάδες. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει 18 εβδομάδες. Οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί, το τι στοιχίζει αυτή η αύξηση από τις 14 εβδομάδες σε 18 εβδομάδες οι μελέτες αποδεικνύουν ότι δεν επιβαρύνει παρά λίγο μόνο τον σχετικό προπολογισμό. 0,02% του ΑΕΠ είναι ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία. 0,02% στη Δανία, τώρα είναι 0,01%, Ισπανία 0,03%. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλή η επιπλέον επιβάρυνση και αν έχουμε μία μητρική, μία άδεια μητρότητας ε, ιδιαίτερα μειωμένη, ίσως, ίσως κάτι που συμβαίνει. Άλλωστε, ίσως η γυναίκα χρειαστεί να ζητήσει και άδεια ε, για ασθένεια της, ε, γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν σε θέση να επανέλθει στην εργασία της και το κόστος του επιπλέον ε, θα ήταν ε, το ίδιο σαν να έμπαινε σπίτι της ε, με την αδιαμητρότητος και ο εργοδότης της δεν θα μπορούσε να οργανωθεί κατάλληλα, να την εγκαταστήσει όπως πρέπει, ενώ αν ζητήσει αδιαμητρότητος αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Ενώ αν τελευταία στιγμή προσθεθεί και άδεια λόγω ασθενείας, τότε μπερδεύονται τα πράγματα. Αυτά λοιπόν αποτελούν λόγους που θα πρέπει να μας σωθούν να νομοθετήσουμε για το πραγματικό όφελος της κοινωνίας και να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά τα 17 τελευταία χρόνια η Ευρώπη και όλος ο κόσμος έχουν αντιμετωπίσει τρομερές αλλαγές. Θα πρέπει να έχουμε και ένα ορίζοντα για το μέλλον να ατενίζουμε και για την ισορροπία της κοινωνίας μας και για την οικογένεια στην Ευρώπη ε, θα πρέπει να προσπαθούμε για το καλό των παιδιών μας. Θα πρέπει να ξοδέψουμε, να δαπανίσουμε κάτι παραπάνω γι' αυτό, παρά να δαπανούμε χρήματα μετά για να πληρώνουμε νοσοκομεία, γιατρούς και φαρμακεία. Εύχομαι να εγκρίνει αυτή την γνωμοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να είναι αντάξιο αυτό που θα βγει του ονόματος του Κοινοβουλίου μας και τίμιο για τους πολίτες μας που τρέχουν ιδιαίτερες προσδοκίες από μας, από τους ευρωβουλευτές. Θέλουμε να έχουμε τη σωστή ενόρεση του μέλλοντος και να αντιμετωπίζουμε τα κύρια προβλήματα που τους απασχολούν. Ίσως σε δύο χρόνια ακόμα θα είναι διαφορετικά τα προβλήματα, αλλά αυτά όμως είναι τα σήμερα αντιμετωπιζόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην εισηγήτριά μας. Πολλές ε, από τις ε, παρεμβάσεις οι οποίες ακούστηκαν αναφέρθηκαν στην ε, γενικότερη συζήτηση και το χορό αυτό άνοιξε ο κύριος Έλμερ εν πάση περιπτώσει ε, φαντάζομαι ότι καλό είναι να ακούμε διαφορετικές γνώμες και να βάλουμε μέσα στην έκθεση όσο γίνεται περισσότερα πράγματα. Όμως διαπιστώνω ότι η κυρία Εστρέλα, εξ ονόματος της Επιτροπής ε, γυναικών το είπε άλλωστε ότι το δημογραφικό ζήτημα θα πρέπει να βαρύνει πολύ στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζομαι το ε, θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν να χαίνομαι δάκρυα επί του δημογραφικού προβλήματος της Ευρώπης και από την άλλη πλευρά να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τι σημαίνει μητρότητα και άδεια μητρότητας ε, στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι και όταν μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία διαρκώς επανέρχονται και τα οποία καταδεικνύουν το... τα περιθώρια που έχουν κάποια δικαιώματα. Δηλαδή υπάρχουν μερικοί που λένε ακούστε κάτι, εμένα σπίτι μου τα πράγματα μια χαρά πάνε και τα κοινωνικά δικαιώματα είναι θαύμα, επομένως δεν με ενδιαφέρει τι μπορεί να πει η Ευρώπη γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι το Κοινοβούλιο έχει ε, διαφορετικό τρόπο συλλογισμού και άλλωστε ε, και ο Μάριο Πόντι ανέλαβε κάποιες ε, υποχρεώσεις και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα γενικά και αυτό να επηρεάσει ακόμα και χώρες οι οποίες θεωρούν ότι είναι υποδειγματικό το δικό του σύστημα. Και μεταξύ άλλων αυτή είναι και η δουλειά του της Επιτροπής. Τελευταία παρατήρηση ε, όσον αφορά την άδεια μητρότητας πατρότητας κατανοώ όλα τα νομικής φύσεως επιχειρήματα τα οποία συνηγορούν υπέρ του να συζητηθεί το θέμα αυτό ε, ε, κάπου αλλού. Όμως από άποψη κοινωνική πιστεύουμε ότι θα πρέπει καλύτερα ε, και προσωπικά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε πιο συνεκτική προσέγγιση και επομένως το θέμα της μητρότητας θα πρέπει να τεθεί σαν ε, θέμα κοινωνικό και σαν, ένα, σαν μια πρόκληση την οποία συνολικά και σφαιρικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή που μιλάμε για έγκυες, για λεχόνες, για γαλουχούσες γυναίκες, ε, ακολουθούμε λοιπόν όλη την πορεία και έχουμε μία συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Εν πάση περιπτώσει, αύριο θα ψηφίσουμε επί των 90 τροπολογιών ε, ή μάλλον θα έπρεπε να πληρώσουμε, να ψηφίσουμε επί των 90 τροπολογιών. Ελπίζω όμως ότι τελικά θα έχουμε μια πιο συνολική ψηφοφορία βάσει των συμβιβαστικών τροπολογιών. Κυρία Εισηγήτρια, τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα το οποίο μόλις ε, μεταφέρατε. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους από όποια πολιτική πτέρυγα ή πολιτική ομάδα και αν προέρχονται. Τους ευχαριστώ για τη συνεργασία η οποία ήδη ήταν πάρα πολύ καλή και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Όσον αφορά τα ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα τα οποία συνδέονται με την ε, κοινωνική αλλά και οικονομική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πω ότι είτε είμαστε γυναίκες είτε είμαστε άντρες βλέπουμε κάθε μέρα ε, τα προβλήματα τα κοινωνικά που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ιδιαίτερα τα προβλήματα που συνδέονται με το θέμα που μας απασχολεί. Ε, Τώρα, όσον αφορά τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, λυπούμε που οι συμβαστικές αυτές τροπολογίες δεν έφτασαν ακόμα σε όλες τις πολιτικές ομάδες, γιατί είχαμε κάποια τεχνικά ε, προβλήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η, συζήτηση Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, ε, θα μπορέσουμε να στείλουμε τις συμβαστικές τροπολογίες σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι όσον αφορά τις ε, αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής μας εδώ, αυτό που είναι σημαντικό είναι να ε, υπογραμμίσουμε τις συνθήκες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, με την προστασία των εργαζομένων γυναικών, ε, για την άδεια, ε, κυρίως δε όσον αφορά την ε, εξολοκλήρου πληρωμένη μητρική άδεια. Θα ήθελα επ' αυτού να καλέσω τους συναδέλφους να σκεφτούν εάν οι δύο ή τέσσερις εβδομάδες οι οποίες φέρονται ως υποχρεωτικές πριν τον τοκετό ε, πρέπει να παραμείνουν ε, υποχρεωτικές. Εγώ είμαι της άποψης ότι οι γυναίκες θα πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιες πώς θέλουν να μοιράσουν την ε, άδεια μητρότητας την οποία δικαιούνται και επομένως να αποφασίσουν και μόνες τους ποια θα είναι, ε, ποιο θα είναι το διάστημα το οποίο θέλουν να σταματήσουν να εργάζονται πριν τον οτοκετό. Σε σχέση με αυτά που είπε η συνάδελφός μου, η Εντίτε Στρέλα, είναι γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση, το δημογραφικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως ε, θα πρέπει να δούμε την μητρότητα εν γέννη σαν ένα ε, κοινωνικό ζήτημα. και επομένως στη γνωμοδότηση εδώ θα πρέπει να είναι σαφής η έννοια της συμφιλίωσης ανάμεσα στην επαγγελματική ε, και προσωπική ζωή όχι μόνο των γυναικών αλλά της οικογένειας γενικότερα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει αναφορά και στην άδεια πατρότητος και όχι μονάχα στην άδεια μητρότητος. Είναι γεγονός ότι εμείς ε, συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή ε, Δικαιωμάτων των ε, Γυναικών και ελπίζομαι ότι εν τέλει θα έχουμε μια γνωμοδότηση η οποία θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κοινωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε αύριο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Γυναικών θα ψηφίσει. Θα δω τα χαρτιά μου και θα σας πω πότε θα ψηφίσει, λέει η Πρόεδρος. Θα εγκρίνει λοιπόν την έκθεση στις 23 Φεβρουαρίου. Και μια και συνεργαζόμαστε άμεσα και στενά, δεν μπορεί να ψηφίσει η Επιτροπή Γυναικών επί των διατάξεων από τον οποίο εμείς έχουμε ήδη ψηφίσει. Αλλά έστω και αν δεν γίνει σεβαστός ο κανένας αυτός, τα μέλη της Επιτροπής ε, μπορεί να επανέλθουν στην Ολομέλεια με τις τροπολογίες που θα έχουν υπερψυφιστεί υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, όπως μας το επιτρέπει άλλωστε ο κανονισμός. Περνάμε επομένω τώρα στο επόμενο σημείο, το σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως, που είναι κομβική σημασία για την οργάνωση των εργασιών μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα πλαίσια μέσα στα οποία οργανώνουμε τη συνάντηση αυτή και το πνεύμα που διέπει τη συνάντηση αυτή. Αντίθετα με την ημερήσια διάταξη που έχει ήδη διανεμηθεί, το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθεί. Επρόκειτο για την ε, συμβολή ε, που θα είχαμε σαν Επιτροπή ε, όσον αφορά ε, την ε, συμβολή μας, ε, λέγω, για την στρατηγική του 2020. Τα πράγματα τώρα έχουν αποσαφινιστεί, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη του Πρόεδρου Στάμπλου, καθώς επίσης και του κυρίου Βαν Ρόμπεϊ. Έχουν ήδη καθοριστεί οι γενικοί προσανατολισμοί και τον Ιούνιο μονάχα θα ε, γίνουν δεκτές οι τελικές διατάξεις, ε, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε σαν Επιτροπή την δυνατότητα αργότερα να ε, πάρουμε θέση όσον αφορά την ουσία ε, αυτής της στρατηγικής. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της θητείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έχει αρχίσει τη δουλειά της και επομένως ε, είμαστε, είναι ακόμα πολύ νωρίς και επομένως στα πλαίσια αυτού του χρονοδιαγράμματος σταματάει η Πρόεδρος. Είναι θεμητό, λέγω, να ακούσουμε τους κοινωνικούς εταίρους, να δούμε τι περιμένουν από αυτήν την ε, θητεία ε, και επομένως να δούμε ποια θα είναι η συμβολή μας όσον αφορά τη στρατηγική 2020 ε, που θα αποτελέσει βεβαίως την σπονδυλική στήλη της μελλοντικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, θα ακούσουμε πρώτα τους κοινωνικούς εταίρους και μετά θα ξεκινήσουμε ε, μια συζήτηση. Ε, θα δώσουμε εδώ δηλαδή το λόγο και στους εκπροσώπους της κοινωνικής ε, πλατφόρμας εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν πράγματα να μας πούν. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο σκέλος ε, δηλαδή στο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με την ε, ε, σύμφωνα το πρόγραμμα που μου έχει προταθεί, θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Τζον Μόνξ ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΤΟΚ. Και θα πρέπει να του ζητήσω να μην ξεπεράσει το οκτάλεπτο. Παρακαλώ κύριε Μόνξ. Ευχαριστώ την Επιτροπή που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να εκφράσω τις θέσεις μας στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Εκ μέρους της ETUC, αλλά πιστεύω και ότι άλλοι συμφωνούν, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια πρωτοφανής ε, διασύνη να περάσει κάτι το οποίο θα μας αποσχολήσει τουλάχιστον για 10 χρόνια ακόμα. Πιστεύω ότι η στρατηγική 2020 σίγουρα θα συμπεριλάβει αυτό το φλέγον θέμα. Θα κάνω λοιπόν μερικές παρατηρήσεις γενικές. Ε, πρώτον, ρωτώ, πέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας. Ε, πολλοί θα πούν ε, ότι βεβαίως πέτυχε. Είναι μια μεγάλη επιτυχία η στρατηγική της Λισαβόνας. Εμείς όμως ήμασταν πολύ πιο επιφυλακτικοί εξ αρχής. Τη ευχηθήκαμε κάθε επιτυχία, είπαμε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να επιτύχει. Αλλά πιστεύω ότι γενικά δεν έχει εκπληρώσει το βασικό της στόχο που, ας μην ξεχνάμε, ήταν να γίνει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο. Και οι λόγοι που δεν πέτυχε το στόχο της είναι προφανείς. Δεδομένου ότι άλλα μέρη του κόσμου αναπτύσσονται ραγδαία και σε μαζική κλίμακα. Πολύ περισσότερο από τη Βόρεια Αμερική και την Δυτική Ευρώπη. Άρα λοιπόν Πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο αυτό που κάνει η Ευρώπη, αλλά και τι κάνουν όλοι οι άλλοι στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Ασφαλώς ε, είχαμε επιφυλάξεις ε, τα τελευταία πέντε χρόνια, από το 2005, για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Τότε η Κομισιόν και το Συμβούλιο είχαν αποφασίσει ότι η ανταγωνιστικότητα θα είναι ο βασικός πυλώνας στον οποίο θα βασιστεί αυτή η στρατηγική. Ο ακρογωνίως λίθος δηλαδή. Εν συνεχεία βεβαίως συμπεριέλαβαν και τα θέματα του περιβάλλοντος στη στρατηγική, αλλά όχι τα κοινωνικά θέματα. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν ήταν επιτυχής αυτή η στρατηγική. Βεβαίως, ορισμένες ε, στρατηγικές ε, στον τομέα της εργασίας ε, προωθήθηκαν σε αρκετά κράτη-μέλη. Δεν λέω, αλλά δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είχε κάποιο συγκλονιστικό, κάποια συγκλονιστική επίπτωση γενικά ε, στην ε, ε, παγκόσμια σκηνή. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε ότι ορισμένες πτυχές ε, της ε, πολιτικής που συζητάμε θα πρέπει να παραμείνουν στα χέρια των κρατών μελών, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι πολλές φορές τα κράτη-μέλη δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους. Η δεύτερη μου παρατήρηση αφορά την προπτική των επομένων 10 ετών. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τα, με τα προσεχή πέντε χρόνια, τα οποία ε, πιστεύω ότι θα τα χαρακτηρίσει η γενική ανάκαμψη της οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μέσα στο πλαίσιο της, ε, της ανάκαμψης πότε θα λήξουν, πότε θα ολοκληρωθούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την οικονομία πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολλά να κάνει αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και ε, της μελλοντικής ανάπταξης. Εάν αυτή τη στιγμή λάβουμε υπόψη ένα 10% ανεργία, δεν πιστεύω ότι έχουμε περιθώριο για μεγάλους ε, ε, για μεγάλη αισιοδοξία και υπερβολικούς ενθουσιασμού ε, μέσα στο πλαίσιο της δεκαετίας. Ε, όχι λοιπόν, ο ουρανό δεν είναι και τόσο γαλανός όσο μας τον περιγράφουν. Στο πλαίσιο λοιπόν των επομένων δέκα ετών και μέσα στην στρατηγική θα πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πολύ περισσότερο σε στρατηγικούς στόχους λείπουν αυτοί οι, κοινωνικοί στόχοι, οι κοινωνική στρατηγική και δεν βρίσκουμε καμία δικαιολογία για την έλλειψη αυτή και πιστεύω ότι αυτό ε, είναι ένα μειονέκτημα και θα πρέπει να το διορθώσουμε. Έχουμε διαπιστώσει στην ε, παρούσα κρίση την αξία της ε, κοινωνικής πτυχής, της κοινωνικής παρέμβασης πάρα πολλές ε, ευρωπαϊκές ε, διαβουλεύσεις έχουν βασιστεί στην κοινωνική σταθερότητα και πάρα πολλές στρατηγικές έχουν στόχο ε, αυτή την σταθερότητα. Σε πολλές χώρες η ανεργία δεν είναι τόσο ψηλή όσο υπήρξε σε προηγούμενες εργασιακές και οικονομικές κρίσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ορισμένες φορές κοινωνικές συνθήκες δεν συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην άμβληση, άμβληση των ε, δυσμενών παραγόντων που έπονται μια τεράστια οικονομικής κρίσης. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να ασχοληθούμε με το καυτό θέμα της αποπληρωμής των δανείων Ποιος θα πληρώσει, το δημόσιο, ο δημόσιος κορβανάς. Θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, τι είδου φόροι, που, σε ποιανού πλάτε θα πέσει αυτή η αύξηση της φορολογίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι γίνονται σοβαρές πολιτικές συζητήσεις για αυτό το θέμα και στα κράτη-μέλη αλλά και γενικά στην Ευρώπη. Γι' αυτό ο πρωταρχικό μας στόχος πρέπει να είναι η προστασία του κοινωνικού συστήματος ε, όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, ιδίως για ομάδες ευάλωτου, για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Θα πρέπει όλοι μας να καταλήξουμε σε μία συμφωνία ότι η κοινωνική πτυχή πρέπει να είναι μία προτεραιότητα στην, ε, στο άμεσο μέλλον αλλά και ε, μέσα στο δεκαετές πρόγραμμα. Όταν μιλάμε για θεμητή αγορά εργασίας, αυτό που έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια είναι η αύξηση της τεράστιας ανισότητας, όπου οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτατα στελέχη των οργανισμών και εταιριών έχουν τεράστιες απολαβές ενώ οι υπόλοιποι πάσχουν και υποφέρουν. Μία τεράστια ψαλίδα λοιπόν έχει ανοίξει όσον αφορά την απασχόληση και τις αμοιβέ. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε δικαιοσύνη και ισότητα στο μέλλον, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ε, εμπειρία μας προηγουμένων ε, περιόδων και όχι να βασιστούμε σε αυτές τις ανισότητες και τις επιρροβολές που σημειώθηκαν τελευταίως. Πιστεύω ότι η συνεργασία με την ETUC είναι σημαντική και χρειαζόμαστε την ενσάρρηση από πλευρά σας για να συνεχίσουμε το έργο μας όσον αφορά την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων, τη βελτίωση της επασχόλησης και των άλλων θεμάτων τα οποία μας απασχολούν. Δεν μας απασχολεί μόνο το δημοσιονομικό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και γενικά ο στόχος των μεγάλων εταιριών. Για ποιανού όφελος λειτουργούν οι εταιρείε, ποιος ωφελείται, ποιος υφίσταται διακρίσεις, είναι μόνο οι μέτοχοι οι οποίοι είναι στόχος ε, των υπέρογκων κερδών που έχουν επιτύχει πολλές εταιρείες. Ε, το συμφέρον των μετόχων πολλές φορές έχει οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές και ακραίες περιπτώσεις όπως είδαμε στις τράπεζες όπου το όλο σύστημα κατέρευσε και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υπέστησαν ε, καρδιακό έμφραγμα. Τι θα κάνουμε λοιπόν για το μέλλον, όχι μόνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και πολύ γενικότερα ε, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Διότι πολλές μεγάλες ε, εταιρείε, ε, επιχειρήσεις ακολουθούν μια ίδια τακτική όπως οι τράπεζες. Βεβαίως ε, είναι υποχρεωμένες να λάβουν υπόψη την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, περιβαλλοντικές ε, ε, παραμέτρους κλπ, ανταγωνιστικότητα και όλα αυτά τα, τα απαραίτητα στοιχεία. Αλλά δεν θέλουμε να ακολουθήσουν μία ακραία πορεία. Αυτές λοιπόν τις παρατηρήσεις είχα πρόεδρε και θα ακούσουμε μεγάλη προσοχή τους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε και σε ευχαριστούμε που σεβαστήκατε το χρόνο μιλίας που είχατε διαθέσεις. Ραλφ Φρέσ από τη ΣΕΠΕ, θα τον παρακαλούσαμε να σεβαστεί και αυτός το χρόνο μιλίας του που έχει στη διάθεσή του. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Είμαι, είναι πρώτη φορά που λαμβάνω μέρος σε, μια τέτοια συζήτηση και είμαι λίγο, έχω λίγο τρακ και ελπίζω να μιλήσω καλά, να μην είμαι υπερβολικά γρήγορος. Όσον αφορά λοιπόν την στρατηγική 2020, η CEEP θεωρείται ως κοινωνικός εταίρος και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή την καρποφόρο συνεργασία με το σώμα σας. Έχουμε πολλές προκλήσεις ενώπιόν μας, καταρχάς ε, ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει να ακολουθούμε μία αξιόπιστη και ρεαλιστική πολιτική για την επόμενη δεκαετία. Η Ευρώπη πρέπει να επιτύχει στην επιλογή μια σωστή στρατηγική. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Κομισιόν να συνεργαστεί και να διαβουλεύεται με του κοινωνικού εταίρου και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι μια πραγματική ευκαιρία ε, επιτυχίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει έναν ε, ε, σημαντικό ρόλο στη διαβούλευση αυτή. Η CEEP έχει εξετάσει με μεγάλη προσοχή τη νέα προσέγγιση, την, τις φρέσκες ιδέες που αναφέρονται για την επόμενη δεκαετία. Συμφωνώ όμως με τον προλαλήσαντα ότι πάρα πολλές ε, κοινωνικές ε, ε, παράμετροι αλλά και άλλοι όπως ο δημόσιος τομέας λείπει τελείω από τις προοπτικές αυτές. Ο δημόσιος τομέας έχει μια εξαιρετική σημασία διότι μπορεί να επιτύχει μια ισορροπία όσον αφορά την, τον τομέα της απασχόλησης σε περίοδους κρίσεων Αντίθετα από, ότι άλλους, από άλλους τομείς, ο δημόσιος τομέας δεν έχει λάβει ε, οικονομικά κίνητρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ένα, ε, είναι ένα τμήμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Δημόσιοι οργανισμοί, δημόσιοι εργοδότες έχουν πολλές φορές ε, ενεργήσει ως μηχανές ανάπτυξης και πρόοδου η ανάκαμψη θα είναι δύσκολη και θα αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις. Οι καινοτομίες, τεχνολογικές ε, καινοτομίες, ε, το περιβάλλον ε, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση ανάμεσα στην καινοτομία και την έρευνα ε, και την ε, απασχόληση. Για, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, συνολική ανταγωνιστικότητα και βεβαίως η γνώση θα παραμείνει στο κέντρο μαζί με την τεχνολογία μια σαφής στρατηγική πρόβλεψης των δεξιοτήτων που θα χρειαστούμε στο μέλλον θα πρέπει να οδηγήσει σε υπηρεσίες οι οποίες θα είναι στελεχωμένες από άτομα καλά εκπαιδευμένα και κατάλληλα άρτια εκπαιδευμένα. Δεν είναι ε, δυνατόν ε, να ε, δυναμητήσουμε την στρατηγική, την γενικότερη στρατηγική μας από τις αλλαγές τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις υποχρεωθήκαμε να, πάρουμε, να κάνουμε λόγω της κρίσης θα πρέπει οπωσδήποτε η αρτιότητα της προετοιμασίας και της γνώσης και της τεχνογνωσίας να συνδυαστεί με έναν ικανό δημόσιο ε, ε, χώρο. Η CEP βεβαίως είναι έτοιμη να παίξει τον ρόλο της και να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας με τρόπο αποτελεσματικό τις επόμενες δεκαετίες. Στρεφόμενος προς τους κοινωνικούς εταίρους και τον ρόλο τους, ε, φυσικά πιστεύουμε ότι θα πρέπει από κοινού να οδηγηθούμε σε μια καλύτερη, επαρκέστερη και οικολογικότερη κοινωνία και οι προτεραιότητες ε, αυτές ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι κοινέ προτεραιότητες οι οποίες ε, θα οδηγήσουν σε μια καλή αγορά εργασίας όπου θα αναγνωρίζονται οι ανάγκες για καλύτερο εργατικό δυναμικό, για αρτιότερο και καλύτερο προετοιμασμένο πλαίσιο έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με τον κοινωνικό αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών. Είναι ένα, ένα από τα πρώτα βήματα που θα μας οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των νέων αναγκών και στην αναγνώριση των δεξιοτήτων που θα χρειάζεται στο μέλλον το εργατικό δυναμικό. Θα αντιμετωπίσουμε επίσης ζητήματα όπως η flexicurity, ε, και ε, όπως η προσαρμογή στην αλλαγή. Στρέφουμε τώρα σε ένα καυτό θέμα, οδηγία χρόνου εργασίας και επ' αυτού πρέπει να πω ότι υψηλής ποιότητος δημόσιος ε, ε, τομέας ε, είναι αυτός ο οποίος έχει και τον χρόνο εργασίας που έχει ήδη αναγνωριστεί σε προηγούμενες οδηγίες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία. Μονάχα η δυνατότητα να θεωρηθεί ο αδρανής χρόνος σαν χρόνος εργασίας ε, θα μας οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό ε, υπολογισμό των όρων ε, εργασίας και νομίζω ότι θα πρέπει προσεκτικά να ακούσουμε τους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά το θέμα αυτό και βεβαίως θα πρέπει να βρεθεί μια δυνατότητα ή τομεακών ή διατομεακών λύσεων τελευταίο ζήτημα. Ο στόχος μας τώρα είναι να διασφαλίσουμε ε, τον εξυγχρονισμό των κοινωνικών υπηρεσιών και ότι ο εξυγχρονισμός αυτός ε, θα οδηγηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως ε, θα πρέπει να συνεχιστεί η, έκθεση η εργασία που ξεκίνησε με την έκθεση Φεραίρο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εξυγχρονιστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και αυτό προς όφελος όλων. Όλοι ε, διαπιστώνουμε αλλαγές στα εθνικά συστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, γνωρίζετε ότι το βάρος, η πίεση των δημοσίων οικονομικών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι ε, μεγάλη και επομένως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρήσουμε και το θέμα των ε, κοινωνικών ταμείων γιατί φυσικά ο αντίκτυπος που έχουν στο ΑΕΠ είναι άμεσος και μεγάλος θα πρέπει να καταρτήσουμε κατάλογο με τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να βοηθηθούμε στο εγχείρημα αυτό και με τούτα τα λίγα ολοκληρώνω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα δώσω τώρα τον, ε, το λόγο στον κύριο Αντρέα Μπενασί, Γενικό Γραμματέα της ε, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα προσκαλέσατε έτσι ώστε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας δώσω πρώτα τρία ε, τρία στοιχεία. 99, 60, 60 είναι αυτά τα τρία στοιχεία κλειδιά τα οποία θα ήθελα να σας αναφέρω. 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλουν κατά 60% ε, στο ΑΕΠ και κατά 60% στην απασχόληση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλο το εύρος των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, δημοσιονομικών κλπ. η ανταλλαγή αυτή απόψεων λαμβάνει χώρα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή ε, όπου όλοι προσπαθούμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να προετοιμάσουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, ε, την EU 2020. Ε, ταυτοποίηση των ε, ε, προκλήσεων. Αυτό είναι πραγματικά από μόνο του μια μεγάλη πρόκληση και ο συνυπολογισμός των δημοσιονομικών περιορισμών, έστω και αν εδώ δεν κάνουμε ακριβώς οικονομική διαβούλευση που θα μας οδηγήσει στην διατύπωση συμπερασμάτων και στην αναγνώριση των παρελθόν των λαθών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες και στο μέλλον για την στρατηγική 2020 έχουμε παρουσιάσει κάποιες προτάσεις όσον αφορά ε, τις αρχές ε, της ε, διακυβέρνησης, της governance και όσον αφορά και την ενεργητική στήριξη των κοινωνικών εταίρων. Ζητούμε συγκεκριμένες και αρκετές βελτιώσεις στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, αν και έχω πάρα πολλά να πω. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο θα πρέπει να ασχοληθεί, να σκύψει με περισσότερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες και συντηρούν και δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας. Ε, γιατί πιστεύουμε ότι πλέον πέρασε ο καιρός που έπρεπε κανείς να βασιστεί και να εστιάσει στις μεγάλες ε, και πολυεθνικές εταιρείες προσβασιμότητα ε, των εταιριών αυτών, των μικρών και μεσαίων εταιριών στις δημόσιες υπηρεσίες ε, γιατί ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα μάλλα εξαρτώνται από ε, τις δημόσιες υπηρεσίες και όσον αφορά τη χρηματοδότηση και όσον αφορά την επιβίωση και όσον αφορά την εκπαίδευσή τους. Όσον αφορά τώρα τον, την αγορά εργασίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικοί σταθεροποιητές της αγοράς εργασίας όσον αφορά, συγγνώμη, γιατί είναι η μεγαλύτερη πηγή, σημαντικό σημαντικότερη πηγή νέων θέσεων εργασίας. Επομένως, η νέα στρατηγική θα πρέπει να ξεπεράσει, να δει παραπέρα από την παρούσα κρίση και εκεί να εστιάσει τι ε, προσπάθειε της. για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, μάκρο και ε, βράχη πρόθεσμες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κινηθούμε προς ε, μια καλύτερη ε, προσέγγιση της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πλέον σε θέση να ενσωματώνει καλύτερα ε, τους εργαζόμενους, να εξισώσει άνδρες και γυναίκες, Τέλος, ε, ε, η ε, συρρήκνωση της αγοράς εργασίας σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν πολύ πιο συγκεκριμένα μέτρα. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι, οφείλουν να έχουν τα δικαιώματά τους, αλλά βεβαίως να ε, δημιουργηθούν και τα κατάλληλα εργαλεία, ας πούμε ένα ή φορολογικό πλαίσιο προσαρμοσμένο δημοσιονομικό ε, ή φορολογικό πλαίσιο το οποίο θα βοηθάει να αποφευθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, μέσω μέτρων και βεβαίως να εξηγιανθούν τα δημόσια οικονομικά από τα οποία μέχρι ένα μεγάλο βαθμό εξαρτώνται οι επιχειρήσεις αυτές η οικονομία, μια οικονομία που βασίζεται στην γνώση χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα περνούν από διαβίου μάθηση, από διαβίου εκπαίδευση και θα εκπαιδεύονται καλύτερα στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς. Be... Ε, τέλος, αλλά όχι Ελλάσσον η επιχει... το επιχειρηματικό πνεύμα θα πρέπει ε, να καλλιεργηθεί και αυτό προς κάθε κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι η πολιτική μικροπίστης, μικροπιστώσεων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Ε, στην στρατηγική όμως του 2020 όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να καλυφθούν με ένα πολύ γενικότερο τρόπο. Ναι, ε, αναφέρθηκα προηγουμένως σε micro credit, σε μικροπιστώσεις. Ε, μάθαμε πολλά πράγματα από την ε, προηγούμενη στρατηγική της ε, Λισαβόνας και ένα από τα μαθήματα που μάθαμε είναι ότι πρέπει να έχουμε πιο στοχευμένες ε, συνεργασίες. Ε, επομένως, πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε όλα να γίνονται με μεγαλύτερη διαφάνεια, να είναι πιο ορατά, να είναι πιο συγκεκριμένα. Να αμβληνθούν οι δυσκολίες μέσω νέων στρατηγικών. Τέλος, εμείς ως ΙΑΠΜΕ είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που κάναμε και στο παρελθόν, δηλαδή να ε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος που θα λάβει το λόγο εδώ στο πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης ε, για την Business Europe δεν μπορεί να είναι ο εισηγητή κανονικά εδώ. Αυτό ο υπεύθυνο της ο Γιούργεν Ρόνεστ θα είναι εδώ από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, και εγώ χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία να ε, μιλήσω ενώπιον της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο διάλογο αυτό. Και η Ένωσή μας, το Business Europe. Η Ευρώπη έχει σημειώσει μεγάλα βήματα ανάπτυξης και εσωτερικά και προς τα έξω, εξωτερικά και πάρα πολλές δυνατότητες καλύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας έχουν αναφανεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε και θα παίξει στο μέλλον ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων. Οι νέες τεχνολογίες, οι περιβαλλοντικές πτυχές, τα προβλήματα τα μεγάλα της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης μας έδειξαν ότι η Ευρώπη πρέπει οπωσδήποτε να εστιάσει την προσοχή της στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην απασχόληση. Έχουμε εδραιώσει συστήματα που ενθαρρύνουν την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Αυτά τα συστήματα όμως τώρα κινδυνεύουν δεν ε, διακυβεύεται πλέον η επιβίωση των ε, συστημάτων ε, κοινωνικών παροχών στην Ευρώπη, της κοινωνικής ευημερία. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε στο μέλλον να αναλάβουμε όλο αυτό το τεράστιο κόστος των κοινωνικών παροχών. Και επίσης ένα μέρος του βάρους αυτού το φορτώνονται και οι επιχειρήσεις. Η καινοτομία και η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι παράγοντες κλειδιά για την ανάπτυξη και πρέπει να δώσουμε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα εκπαίδευσης ε, στις δεξιότητες που χρειάζονται στο μέλλον. Οι προτεραιότητες που έχει δώσει η Κομισιό σε αυτό τον τομέα είναι φιλόδοξες, αλλά πιστεύω ότι είναι σωστές. Ε, πρέπει να μετακινηθούμε σε οικονομίες οι οποίες είναι πολύ πιο πράσινες, είναι οικονομικά βιώσιμες, πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαβίου εκπαίδευση των εργαζομένων και ιδίως των ανθρώπων που εγκαταλείπουν ε, τη σχολική εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία. Η Επιτροπή ε, Παιδείας πιστεύω ότι έχει επικεντρώσει την προσοχή σε αυτό το θέμα της διαρκούς εκπαίδευσης. 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα βγουν από την αγορά εργασίας τα επόμενα 40 χρόνια. Είναι ενδεχόμενο οι ρυθμοί ανάπτυξης να κοπούν στο, στο ίμιση, να μειωθούν κατά το ίμιση. Αυτά τα 40 εκατομμύρια θα ενταχθούν στο πλαίσιο συνταξιοδότησης και καταλαβαίνετε βεβαίως ότι χρειάζεται πολύ σοβαρή μελέτη της, ε, του συνταξιοδοτικού πλαισίου και του βάρους αυτού στα ευρωπαϊκά κράτη. Ο επιχειρηματικό κόσμος πιστεύει ότι πρέπει να επικεντρώσετε την προσοχή σας, εσείς δηλαδή, εδώ στο Ευρωπαϊκό Σώμα, στα εξής. Πρώτον, σύγκληση και οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς ε, είναι και ο στόχος ε, της ε, κοινή αγοράς, της εσωτερικής αγοράς. Μία οικονομική σύγκληση που να οδηγεί στην ανάπτυξη. Η στρατηγική 2020 θα επιτύχει μόνο εάν τα κράτη-μέλη ενθαρρυνθούν να επιβάλλουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στην προσπάθεια αυτή και να ενθερρύνει την ε, επαγγελματική εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων. Πρέπει λοιπόν και εδώ να εφαρμόσουμε τις αρχές της ευελιξίας και της ασφάλειας, το flexicurity όπως λέμε στα αγγλικά, και να το ενσωματώσουμε ε, ώστε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους να παραμείνουν στην αγορά εργασία. Πρέπει επίσης να τους δώσουμε κίνητρα αναζήτησης άλλης εργασίας, σε περίπτωση που έχουν χάσει τη δουλειά τους, και συνεχούς εκπαίδευσης, περαιτέρω εκπαίδευσης. Πάνω από 70 οδηγίες έχει ο τομέας εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και ο θεμέλιος, ε, οι πυλώνες της πολιτικής αυτής ε, εξασφαλίζονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη περισσότερης νομοθεσίας και ενός ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω, εμείς πιστεύουμε, ότι θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην καλύτερη και πληρέστερη εφαρμογή των διατάξεων που ήδη περιέχονται σε αυτό το πλαίσιο. Τα τελευταία δέκα χρόνια και έχουν σημειωθεί πάρα πολλές αλλαγές και αυτές έχουν ληφθεί υπόψη στην πολιτική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία πρώτον στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις ώρες εργασίας πρέπει να ρυθμίσουμε καλύτερα το όλο θέμα των ορών εργασίας. Η οδηγία του 1993 ε, δεν αντανακλά πλέον τη σημερινή πραγματικότητα της Ευρώπης και δεν αντανακλά τις αλλαγές που έχουν γίνει στον χώρο εργασίας και την απαραίτητη ευελιξία η οποία απαιτείται συζήτηση για την τυχόν αναθεώρηση της οδηγίας αυτής πέρσι δείχνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε τον τομέα των υπηρεσιών, να τον διευρύνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας προστασία στους εργαζόμενους. Η εφαρμογή του πλαισίου αυτού στα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιωθεί, αλλά δεν χρειάζεται περαιτέρω ε, νομοθεσία πρέπει να διορθώσουμε τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει αυτές τις ανάγκες. Έχουμε αναθεωρήσει, αναθεωρήσει ε, την Συμφωνία Πλαίσιο για τη γονική άδεια. Έχουμε επίσης ε, προσφέρει τις, ε, τις απόψεις μας, τις συμβουλές μας ε, στο, στην αγορά εργασία και τη διαμόρφωσή της στο μέλλον και τώρα εργαζόμαστε πάνω σε μια κοινή σύσταση για τη στρατηγική 2020. Έχουμε επίσης μελετήσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τους ερχόμενους μήνες θα παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη μας έκθεση. Οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι έχουν μόλις ολοκληρώσει τη μελέτη τους για το τι χρειάζεται στην αγορά εργασία και θα παρουσιαστεί το Μάρτιο του 2010. Προσπάθησα να σας ε, παρουσιάσω τις προσδοκίες μας που έχουμε για τα επόμενα 10 χρόνια. Όμως ε, δεν ε, πρέπει να παραλείψω και τις μεγάλες ανησυχίες, τις άμεσες της οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν ορισμένα σημάδια ανάπτυξης, αυτή, ε, ε, ανάκαμψη συγγνώμη, αυτή τη στιγμή. Όμως η κατάσταση στην αγορά εργασίας δεν θα βελτιωθεί σύντομα. Δεν έχουμε σημάδια άμεσης βελτίωσης. Ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία έχουν καταφέρει να περάσουν την κρίση αυτή πιο ήπια. Άλλες χώρες τις έχει χτυπήσει η ανεργία πολύ σκληρότερα. Όμως όλοι αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε. Ο αγώνας για την επιβίωση είναι κοινό χαρακτηριστικό στην Ευρώπη. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι πολιτικές οι οποίες θα παρεμποδίσουν την αύξηση σε χρηματοδοτικές πηγές ή που θα αυξήσουν το κόστος εργασίας. Προς Θεού δεν χρειάζονται τέτοιες πολιτικές. Είναι λοιπόν ε, ε, απολύτω αναγκαίο να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την κατάσταση στην αγορά εργασία. Ευχαριστούμε τους τέσσερις συγγετές μας οι οποίοι ξεκίνησαν και την όλη, το όλο θέμα. Έχω τον κατάλογο μιλητών, θα κλείσει 2,3 ομιλητές, αλλά τελειώσαμε, δεν δεχόμαστε άλλους. 11 έχουμε ήδη. Και δυστυχώς δύο λεπτά ο καθένας και Σέρκας δύο λεπτά και Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε. Όλοι έχουμε συνέστηση ότι ξεκινάμε μια νέα φάση, νέες συνθήκες, νέα στρατηγική, νέα επιτροπή, νέο το κοινοβούλιο νέα φάση λοιπόν θα έπρεπε να κάνουμε σαν πρώτο όχι να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Το 2010 έτσι θα ολοκληρωθεί με διάφορες εκλογές και θα δούμε ότι η Ευρώπη υποφέρει από πολλές κρίσεις και αν είμαστε ικανοί θα δούμε ότι δεν είναι μόνο οικονομική κρίση. Σίγουρα είναι και οικονομική κρίση, αλλά είναι και κρίση αξιών κοινωνίας ε, μας σαν ε, και του ευρωπαϊκού του σχεδίου αυτού καθ' αυτού που δεν είναι μόνο οικονομικό σχέδιο. Και το μεγαλύτερο λάθος αυτά τα χρόνια ήταν ε, την Ευρώπη να την περίσουμε μόνο στην οικονομική της πτυχή και να ξεχνάμε τους εργαζόμενους, τους πολίτες μας, τις επιχειρήσεις μας, τις περισσότερες επιχειρήσεις, αυτό τον ιστό τον παραγωγικό στην Ευρώπη που καταστράφηκε από μια αγορά που τρελάθηκε χωρίς καμία ρύθμιση και το μεγαλύτερο κέρδος που επιδιώκει ο καθένας, αυτό καταστρέφει τα πάντα, την κοινωνία, την οικονομία, τις ίδιες επιχειρήσεις, μπούμεραγκα, αυτό αντιμετωπίζουμε και για να δούμε, έχουμε νέα περίοδο τώρα, δεν ξέρω αν οι κοινωνικοί εταίροι θα καταβάλουν την προσπάθεια πέρα από τους πολιτικούς ε, να συνεργαστείτε, να δούμε, να δούμε αυτές τις παλιές ουτοπίες ίσως 40-50, ε, μια νέα Ευρώπη για τους πολίτες, ε, μια πορεία να αλλάξει η κατάσταση στα κοινωνικά και στα οικονομικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει πρόεδρος. Δυστυχώς, ε, εντάξει, κάτι που δεν θα βοηθήσει τον με τον άλλο θα κάνω, αλλά για να μπορέσει ο καθένας ε, να λάβει το λόγο και μετά να δούμε και τους συζητητές μας πώς θα απαντήσουν. Ευχαριστώ, λέει κυρία μαρέν Ευχαριστούμε για την οργάνωση ακρόαση αυτή με του ε, μα για την όλη εξέλιξη τη στρατηγική. Να μην επανέλθω τώρα σε θέματα που ο κ. Σέρκας ε, είπε για την κρίση και για το νόημα που έχει αυτή η κρίση. Θα ήθελα τάχιστα να θίξω τέσσερα σημεία. Το πρώτο σημείο ποιο είναι. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Η κοινωνία που την, όπως την επιθυμούμε στα πλαίσια της της Λισαβόνας να είναι μια κοινωνία που θα πετύχει, να είναι μια κοινωνία γνώσης, ε, και θα ήθελα τώρα να μιλάμε για κοινωνία της επιτυχίας. Τι σημαίνει επιτυγχάνω και να περιλαμβάνω καινοτόμα στοιχεία, αλλά ο καθένα να μπορεί να έχει τη θέση του στον επαγγελματικό κόσμο, γιατί ακριβώ η ένταξη κοινωνική από αυτά βγαίνει. Επαγγελματική κοινωνική ένταξη. Αυτή θα είναι μια επιτυχημένη κοινωνία. Και δεν μπορούμε να κεστούμε μόνο σε λόγια σε αυτά. Δεύτερο σημείο. Οι υπηρεσίε του δημοσίου. Οι υπηρεσίε θα πρέπει να αποτελούν κινητήρια δύναμη στην όλη ανάπτυξη, εξέλιξη τη κοινωνία όπω την επιθυμούμε στην Ευρώπη. Τρίτο σημείο. αυτή την πετυχημένη κοινωνία δεν θα την έχουμε εάν δεν περάσουμε μέσα από μια νέα ένα νέο διακυβέρνηση για να πετύχουμε και τη στρατηγική Λισαβόνα, όπως είπαν και αρκετοί ομιλητέ, Αναρωτιόμαστε πώς θα πετύχει αυτή η στρατηγική της ε, θα πετύχει μόνο όταν θα μπορούμε οι ίδιοι μαζί μα ε, να έχουμε μια ενόραση, όχι εθνική αλλά και περιφερειακή. Η κοινωνία η πετυχημένη θα περάσει και μέσω μια διεθνού αλληλεγγύη. Σα ευχαριστούμε. Σάντζο Κομφεράτη και μετά το Μασμένου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας Ποια θα είναι η άποψή τους ε, για διάφορα προβλήματα που τόνισαν ε, οι ίδιοι, αλλά δεν έφτασαν ε, σε τελικά συμπεράσματα αυτά τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2020 δηλαδή. Εκεί όλοι συμφωνούν και οι οικονομολόγοι που ασχολήθηκαν ότι θα έχουμε μακράς διαρκείας ανεργία, λόγω της αγοράς εργασίας και των δυσκολιών της και ακόμα μια πολύ μα πολύ αργή ανάπτυξη και οι πόροι για τις δημόσιες δαπάνες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές για και το χρονικό διάστημα. Εδώ, από αυτά τα στενά, θα πρέπει να πετύχουμε με τις ε, χαμηλότερες κοινωνικές ε, θυσίες αυτό το θέμα και εδώ, όταν θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε πάλι για ωράριο εργασίας, θα δούμε και την διάρκεια το χρόνο εργασίας και όχι μόνο την όλη ευκαμψία και ευληγησία χωρίς ανακατανομή της υπάρχουσας του υπάρχοντος όγκου εργασίας δύσκολα οι επόμενες δεκαετίες όσον αφορά την απασχόληση θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης εύκολης ε, ε, από την κοινωνία μας και ακόμα πρότυπα πρότυπα που θα προσδιοριστούν ώστε να μην ξαναπέσουμε και πάλι σε τρομερά προβλήματα στη δημόσια δαπάνη επίσης και τις συνδικαλιστικές σχέσεις και εκείνε θα πρέπει να εξεταστούν και να δούμε λεπτομερώς για να δούμε και κύριες γραμμές συνεννόησης για μικρότερες πιθανότητε σύραξης και περισσότερη συνεργασία και ε, χαμηλότερη ένταση κοινωνική, μη διαχειριζόμενη σωστά, επειδή θα υπάρχουν τα μέσα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τόμας Μαν και Κέζιν Λαμπέρτ στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ομιλητές. Έχω τρεις ερωτήσεις. Είχαμε μία πολύ καλή έκθεση για το flexicurity, ευελιξία και ασφάλεια από τον Όλε Κρίστεν που είναι εδώ. Από τη μία μεριά έχουμε την ευελιξία, από την άλλη την ασφάλεια, επίκεντρο αυτής της έκθεσης. Άκουσα ότι δεν υπάρχει επαρκής κοινωνική ασφάλεια. Ε, μήπως αυτή η παρατήρηση οφείλεται στο ότι η Κομισιόν έχει μόνο ένα μικρό κεφάλαιο αφιερώσει σε αυτό το θέμα. Τι πιστεύετε, απευθύνουμε στο πάνελ. Και ε, πρέπει επίσης να αναφερόμαστε σε στρατηγικές εισόδου στην αγορά εργασίας, αλλά και σε στρατηγικές παραμονής. Στην χώρα μου έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη χρηματοδότηση της μερικής απασχόλησης για ε, περιορισμένο σύντομο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους όταν η προσωρινή τους απασχόληση τελειώσει. Πρέπει να υπάρχουν άλλες ε, επιλογές παραμονής στον τομέα της εργασίας. Και ένα θέμα δεν το οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου, τι γίνεται με τη μαύρη αγορά εργασίας. Αυτός ο τομέας επιβαρύνει, ζημιώνει τους εργοδότες, όχι αυτούς τους εργαζόμενους, τι δυνατότητα έχουμε λοιπόν να περιορίσουμε ή να ε, πολεμήσουμε τη μαύρη αργορά εργασίας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και την επιβίωση των νομίμων, νομίμως εργαζομένων. Και μία ερώτηση για τον κύριο Ρόνερτ. Ανέφερε την οικονομία πολλές φορές και την οικονομική ανάπτυξη και είπε ότι χρειαζόμαστε και περισσότερη ανάπτυξη στην ψηφιακή τεχνολογία. Ε, μήπως αυτό είναι λεπτομέρεια. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε είναι ομάδες εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν αρμονικά μεταξύ τους για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εντελώς καινούργια αντίληψη, συλλογική, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Όπως ακριβώς το κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπληρώνει η Πρόεδρος. Τζιν Λάμπαρτ και μετά ο κ. Πουπάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως ακούσαμε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, είτε ήταν σωστά είτε επικριτικά όσον αφορά τον ρόλο της δημόσιας ε, του, του, του, του δημόσιου τομέα που είναι σημαντικός. Τώρα όσον αφορά την στρατηγική 2020 ε, διαπιστώνουμε ότι αυτή ε, δεν είναι πλήρως εναρμονισμένη με άλλες στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτές τις στρατηγικές που αφορούν την Ένδια, δεν κάνουμε πολύ μεγάλη πρόοδο στο θέμα αυτό. Τώρα ασχολούμαστε και με στρατηγική αηφόρου ανάπτυξης. Το κλίμα αναφέρθηκε από πολλούς και επίσης βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ φτωχών και πλουσίων και το κοινωνικό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτής της ε, διάστασης. Ε, αυτή η διασύνδεση ανάπτυξης ε, και απασχόλησης ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η στρατηγική 2020 κάνει πολύ λόγο για ανάπτυξη, χωρίς όμως να δίνονται πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό. Δίνεται μάλλον η αίσθηση ότι η ανάπτυξη αυτόματα σημαίνει και αύξηση της απασχόλησης. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε είτε ε, την ανάπτυξη είτε τις θέσεις εργασίας και να δούμε ποια ακριβώς είναι η διασύνδεση μεταξύ των δύο. Επίσης, αυτή η στρατηγική 2020 πώς μπορεί να ενταχθεί στις νέες ε, παγκόσμιες προκλήσεις ε, τις οποίες εσείς ακροθυγώς αναφέρατε. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε από την κοινωνική πολιτική, από το περιβάλλον, από όλες τις πολιτικές, πώς ακριβώς μπορούμε να εντάξουμε, να ενσωματώσουμε τις πολιτικές αυτές στη στρατηγική 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πουπάκης και μετά ο κύριος Μαύρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και η μεταξέλιξή της σε κρίση απασχόλησης ανέδειξαν με επώδυνο τρόπο την αδυναμία της στρατηγικής Λισαβόνας 2010 και επέτειναν την ανάγκη για να περθούν μέτρα να υπάρξουν κοινωνικέ μεταρρυθμίσει. Βλέποντα την πραγματικότητα σήμερα, έχουμε ένα ιδιαίτερα ποσοστό ψηλού ανεργία στα κράτη-μέλη που δεν προβλέπεται να μειωθούν τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια. 19 εκατομμύρια φτωχού εργαζόμενου, αποτέλεσμα τη ραγδαία και χωρί θεσμικό πλαίσιο επέκταση του θεσμού των ευέλικτων μορφών εργασία, με 80 εκατομμύρια συμπολίτε να διαβιούν κάτω από τα όρια τη φτώχεια, έτσι συνθέτουν ένα σκηνικό απορρίθμιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Εδώ συμβάλλουν και δυστυχώ και έντονε διαφοροποίησει στα εθνικά εργασιακά καθεστώτα και νομοθεσία των κρατομελών, καθώ και μία επικύρωση από πάρα πολλά κράτη-μέλη των διεθνών συμβάσεων εργασία, έχοντα δημιουργήσει έντονο θεσμικό έλλειμμα, με αποτέλεσμα να φύγεται το δικαίωμα στην εργασία με αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη δίκαια με βίη, στη δικαστική ελευθερία, η αποτελεσματική πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και στον έλεγχο τη στήριξη εργατική νομοθεσία. Έτσι χρειάζονται μεταρρυθμίσει. Είναι εντελώ απαραίτητε. Όμω οι όποιε αναγκαίε μεταρρυθμίσει δεν μπορούν και δεν πρέπει να επιβληθούν από πάνω. Απαιτείται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των εθνικών κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, τη οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, με τη δημιουργία ενό νέου θεσμικού πλαισίου ουσιαστική συμμετοχή του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένω, το πλαίσιο κατάρτιση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και με υπευθυνότητα αυτές τις εργασιακέ προκλήσεις για την απεναξέταση και βελτίωση της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και τη συνεργασία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών να διασφαλιστεί και να ενδυναμωθεί η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης που σε αυτή την περίοδο της κρίσης δυστυχώς βρίσκεται σε κίνδυνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και μετά ερωτήσεις. Λοιπόν, σχετικά με τους κοινωνικούς εταίρους και τις παρεμβάσεις, αυτή η στρατηγική 2020 έχει ένα αδύναμο σημείο. Δεν υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα στοιχεία και είναι πολύ γενική αυτή η στρατηγική. Να πω μερικά πράγματα που αισθάνομαι την έλλειψή τους. Παλιότερα με τη στρατηγική της Δισαβόνας είχαμε αναφερθεί ιδιαίτερα σε διάφορα στοιχεία στα οποία τώρα δεν αναφερόμαστε. Πάνω απ' όλα την κοινωνική συνοχή. Υπάρχουν πολλές διαφορές στην κοινωνία μας. Και ακόμα στο έγγραφο αυτό κυρίως πρόκειται για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα εξασφαλίσουμε τη ροή υπηρεσιών, διαφάνεια διαφόρων συστημάτων και πώς γενικά θα εγγυηθούμε μια ανάπτυξη, μια, ένα υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης. Αγαπητοί εισηγητές, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας σε αυτά. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τη στρατηγική απασχόλησης και εκεί συμφωνούμε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και επίσης συμφωνούμε για το ρόλο που παίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι σημαντικότατος. Και ακόμα ο νέος τρόπος ε, διαχείρισης ε, δεν ξέρουμε όμως λεπτομέρειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρμοδιότητες επ' αυτού. Το Συμβούλιο θα είναι κανονικά η κινητήριος δύναμη στην αλλαγή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυστυχώ δεν συμμετέχει παρόλο που λειτουργούμε από την 1η Δεκεμβρίου που μας πέρασε με διαφορετικό τρόπο αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τα πλαίσια μα. Ναι και εγώ ίδια θα λάβα το λόγο και μετά ο σε Εδώ θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου γιατί η Επιτροπή έστω και αν δεν έχουμε τη νέα σύνθεση της ακόμα στις διαπραγματεύσεις αυτές ε, και το κείμενο που είναι διαθετική σημασία, δεν ξέρω, δεν έχει καταλήξει κάπου. Θα πρέπει να δούμε για τις ηγητέ. Για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού είναι από του λόγου αποτυχία τη θετική λύσης αγορά. Τι θα κάνουμε στα πλαίσια της 2020, 2020 και ακόμα κάτι. Πέστε μου κάτι. Τρία σημεία που σα φαίνονται ότι είναι σημαντικά από τη στιγμή που θα δούμε αυτό το θέμα τη διαχείριση, όπω είπε ο Τζον Μόγκ και που κάτι την απόψή μου έχει είναι ουσιώδες για να δούμε προς τα που θα στραφεί αυτή η πραγματικότητα όσον αφορά τη βάση λειτουργίας των επιχειρήσεών μας. Στα πλαίσια αυτά, τι φρονείτε εσείς ε, επειδή υπάρχουν επικουρικά ταμεία ασφάλισης, ε, είναι σημαντικό αυτό, είτε μπορούμε να το παραβλέψουμε, δεν νομίζω. Στα πλαίσια δε τα ίδια, τι θεωρείτε επειδή πολλές φορές αναφέρομαι στο ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά πολλοί κανεί δεν το κοίταξε κατάματα, δηλαδή αν χρειάζεται ή όχι μια οδηγία πλαίσιο. Εδώ εξαντλείται το θέμα αυτό από τη στιγμή που ισχύει πια η στρατηγική τη Αβώνας, είτε θα πρέπει να το επαναξεταστεί. Αυτά σύντομα, σύντομα τηλεγραφικά. Δεν ξέρω αν θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε σε όλα. Αυτά πάντως εμένα με απασχολούν. Φρανσουάς ε, Καστέξ ε, και μετά Ελίζαβετ. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ τάχιστα να αναφερθώ στην πρόταση της Επιτροπής και δύο-τρεις ερωτήσεις να υποβάλω στους εισηγητές. Τρεις ρωτησεις να υποβαλω στους εισηγητες τρεις παρατηρησεις για το κείμενο της Επιτροπής. Ε, δεν έχουμε την ανάλυση παλιότερα τη στρατηγική τη Σαββόνα. Όταν προτείνεται μια νέα στρατηγική αντί για μια άλλη, αυτό πρέπει να γίνει, τουλάχιστον να δούμε τι γίνεται σε αυτό. Είδαμε διάφορου στόχου, απασχόληση, το απασχόληση των γυναικών, ηλικιωμένων ατόμων, ε, νέων και παιδιών, φροντίδα, δεν έχουμε τίποτα εκεί, ούτε επίσης για την κρίση την κοινωνική, που, για τη φτώχεια, για τους άνεργους, για τον κοινωνικό αποκλεισμό, ούτε και ενεργός πολιτική ενσωματωμένη εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε αυτό το ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Πέρα από αυτή λειτουργούμε. Εδώ μιλάμε μόνο για ε, πώς θα επηρεαστούν τα πράγματα χωρίς να μιλήσουμε ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο ούτε σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Εδώ λοιπόν ε, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν φιλοδοξίες όσον αφορά τα μέσα και για τους συγητές μας. Ο κύριος Μόγκ έθεσε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, θα ήθελα να μας το αναπτύξει. Λέει, ποιο θα σηκώσει το βάρο αυτή τη συμπερίληψη τη κοινωνική. Δεν υπάρχει τίποτα στο κείμενο αυτό. Θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει με τα οικονομικά μέσα, ποιο θα υπομειστεί ακριβώ αυτόν τον τομέα την ανακατανομή του πλούτου. Okay. Όταν μιλάτε για τις μας υπηρεσίες και πώς θα επαναλειτουργήσουν σωστά, εμείς όλοι είμαστε υπέρ αυτής της δημόσιας υπηρεσίας. Ε, η επανεκκίνησή τους είναι κάτι σημαντικό. Σας παρακαλούμε μήπως θα μπορούσατε να μας αναπτύξετε δηλαδή αυτή. Για τον κύριο Ρόνεστ ένα ερώτημα. Λέτε ότι θα έχουμε 40 εκατομμύρια Ευρωπαίους που θα... δεν θα εργάζονται πλέον. Ε, υπάρχει ένα έλλειμμα λοιπόν εργατικών χεριών. Το πρώτο, τι λέτε, πρώτη, τι είναι περισσότερη χρόνος ε, εργασίας ε, και όχι για τους υπόλοιπους να μπορούν να εργαστούν οι γυναίκες το κατάλληλο και αντί να λέτε περισσότερο χρόνος εργασίας για αυτούς περισσότερα χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Από ό,τι άκουσα γενικά, δεν πιστεύετε ότι η στρατηγική της Λισαβόνας θα την επιτυχημένη. Ε, πολλοί θα ε, συμφωνούσαν μαζί σας ότι δεν πέτυχε τους στόχους της. Ιδιαίτερα στο θέμα της, του κοινωνικού αποκλεισμού ε, δεν πέτυχε. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς πιστεύετε ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να βοηθήσουν σε, σε αυτή την έλλειψη. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που δημιουργούν διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Επίσης, σχετικά με την υλοποίηση, την εφαρμογή των οδηγιών που είπατε πρέπει να βελτιωθεί. Τι μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να κάνουν για να βοηθήσουν την πλήρη και καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών. Υπάρχει κάποιες, υπάρχουν συλλογικές δραστηριότητες που μπορούμε να αναλάβουμε για να βοηθήσουμε θα θέλαμε εμείς ε, ως Επιτροπή Επασχόλησης να ακούσουμε από εσά αν το θεωρείτε αυτό το θέμα ως θέμα προτεραιότητας. Επίσης, ένας από εσά ανέφερε την τομεακή προσέγγιση της Κομισιόν. Πιστεύετε ότι ε, ο τομέας της υγείας, παραδείγματος χάρη, από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να βελτιώσουμε την απασχόληση ή όλοι πιστεύετε ότι αν ασχοληθούμε με τον τομέα της υγείας ενδέχεται να καταλήξουμε σε μερική συμφωνία αλλά θα αγνοήσουμε τους υπόλοιπους τομείς. Ήταν καλή ιδέα δηλαδή. Η κυρία Φιγκερέρο και μετά η κυρία Σρέντερ. Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ όταν ζητείτε να προσέξουμε ακριβώς τη δίκη που η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε για κοινή συζήτηση και διαβούλευση και η οποία και ολοκληρώθηκε 15 Ιανουαρίου, λίγο πριν από την εγκατάσταση της νέας επιτροπής, κάτι που δεν έγινε όμως και αυτό δεν στέκει, δεν συνάντη με τα υπόλοιπα δεν έχουμε ούτε καν ανάλυση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πριν από δέκα χρόνια μιλούσαμε για πλήρη απασχόληση. Λέγαμε να μειωθεί η φτώχεια. Λέγαμε ότι έπρεπε να υπάρξει κοινωνική συνοχή και αύξηση το ΕΠ κατά 3%. 3%. Τώρα τα τελευταία στοιχεία της Eurostat το 17% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτωχός πληθυσμός. Είναι 85 εκατομμύρια άτομα που ζουν φτωχά. Και αυτό τέλη του 2008. Τώρα με την κρίση θα έχουμε ακόμα περισσότερους. Πάνω από 24 εκατομμύρια ανέργους έχουμε οι νέοι είναι το 21% των ανέργων και όσοι εργάζονται είναι σε κίνδυνο αυτή η θέση εργασία τους και κακοπληρώνονται. Όλα αυτά θα πρέπει να τα παραδεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τρομερό το κενό και προκλήθηκε από τις πολιτικές της που δεν ήταν σύμφωνες με τις προαναγγελθήσεις πολιτικές που θα έπρεπε να ασκηθούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν νομίζω ότι λείπει ο σχετικός απολογισμός και ακούμε ανήσυχα να τονίζονται διάφορες προτάσεις. Ακούγεται ότι μεγαλύτερο ωράριο εργασία. Τι θέλουμε, με αυτά τα προβλήματα, ακόμα περισσότερες ώρες εργασία παρόλο που άνεργοι νέοι υπάρχουν. Στρέτερ. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται διερμηνία στα δανέζικα, γι' αυτό θα μιλήσω αγγλικά. Ε, η κυρία Σρόντερ όμως είπαμε πρώτα. Α, πρώτα η κυρία Σρόντερ και μετά. Ναι, εντάξει. Κυρία Σρόντερ λοιπόν. Ευχαριστώ, θα είναι πολύ σύντομη. Πρώτον, με εντυπωσίαση η ευγένειά σας προς την Κομισιόν. Εδώ έχουμε μία στρατηγική 10 ετών και αυτό που βλέπουμε δεν αξίζει την αξία του χαρτιού που έχει γραφτεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν να εκφράσουμε ξεκάθαρα την άποψή μας. Όπως είδαμε, ε, ε, υποχρεώνονται οι επίτροποι να ε, εκδώσουν αυτήν τη στρατηγική για να δείξουν στον κόσμο ποια είναι η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πράγμα δεν ε, πέτυχε το στόχο του. Δεν τα κατάφεραν. Θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να πούμε, να ξέρουμε εσείς πώς φαντάζεστε τη στρατηγική της επόμενης δεκαετίας, τη μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να κάνουμε σημαντικές και ριζικές διορθώσεις. Δεύτερον, υποτίθεται ότι η στρατηγική αυτή λέει ότι θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μια πιο οικολογική οικονομία, πράσινη οικονομία. Ε, εντάξει, η ιδέα είναι σωστή, αλλά χρειαζόμαστε και την ε, εμπειρογνωμοσύνη, το know-how γι' αυτό. Από πού θα βρούμε τους ειδικού και τους εμπειρογνώμονες ε, να κάνουν αυτή τη μετάβαση. Παρακαλώ λοιπόν να ληφθεί υπόψη και αυτό το θέμα της ανάγκης εμπειρογνωμόνων. Εν συνεχεία αναφέρει αυτή την ε, εκστρατεία εκ, ε, Για ποιον, για ποιον προορίζεται αυτή η εκστρατεία δεν έχουμε καμία συγκριτική πολιτική. Συμφωνούμε όλοι στο στόχο αυτό. Θα με ενδιαφέρε λοιπόν ιδιαίτερα να ακούσω από εσά τι υποχρεώσεις πρέπει να έχουν οι εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αυτές οι γενικότητες και με τι, τι κονδύλια χρειάζονται για να εφαρμοστούν αυτές οι γενικότητες που αφορά αυτό το χαρτί που λέει στρατηγική 2020. Τώρα η κυρία Τουρίνεν. Ευχαριστώ. Αυτό μου εκπλήσει όταν ακούω όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι σε αυτές τις στρατηγικές ε, γίνεται μια προσπάθεια οικοδόμησης της αλήθειας. Ε, είπατε πολλοί από εσά ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα ασφάλισης και αυτό είναι αλήθεια. Ε, αλλά αυτό είναι η εκδοχή μίας, μία εκδοχή μίας αλήθειας. Ε, η υπόλοιπη αλήθεια είναι τι γίνεται με όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση, εκπαίδευσή τους και που με κάποιο τρόπο θα πρέπει να μπουν σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να μην δεχόμαστε κάποιες ε, αλήθειες ή κάποιες πλευρές αλήθειας που λένε ας πούμε, ότι πρέπει να είμαστε άμεσα ανταγωνιστικοί κτλ. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση οδηγείται προς πολλές ε, κατευθύνσεις και άλλωστε έτσι πρέπει να είναι γιατί η στρατηγική αυτή είναι πολύ ευρεία και επομένως θα πρέπει ε, να ε, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και επομένως να μπούμε σε λεπτομέρειες. Να μπούμε κάτω αν θέλετε από τις επικεφαλίδες πράσινη οικονομία, ε, κοινωνία κτλ. Να, να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα απτά απαντήματα, γιατί, συγγνώμη, με συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Γιατί ξέρετε, δεν θα καταφέρουμε τελικά να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων και να αντιμετωπίσουμε ας πούμε την Ινδία ή την Κίνα. Γιατί και εκείνοι προχωρούν όσον αφορά την εκπαίδευση ε, και πολλά άλλα πράγματα. Η Ισπανική Προεδρία ε, μας ε, παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ένα πρόγραμμα βασισμένο στην ισχυρή διακυβέρνηση, governance. Τι γίνεται όμως, ποια είναι τα εργαλεία τα οποία έχουμε, ποια είναι τα εργαλεία τα οποία μας, δίνει, ε, μας δίνουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να βάλουμε έτσι ώστε να αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή η πράσινη οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ακούσατε τα μελήματα όλων των ε, ε, ε, αγοριτών, όλων των μελών του Κοινοβουλίου και αυτό είναι θετικό, αλλά υπάρχει και αρνητικό, έχετε μονάχα τέσσερα λεπτάκια έτσι ώστε να απαντήσετε. Αλλά όμως μην πέσετε στην παγίδα να μην μας πείτε τίποτα, δηλαδή να είσαστε πολύ γενικόλογοι ε, με το πρόσχημα δεν έχω χρόνο να απαντήσω. Διαλέξτε ένα θέμα αν είναι ανάγκη και απαντήστε πραγματικά ουσιαστικά σε αυτό το ένα θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με ένα με την ερώτηση κυρίας Λάμπερτς. Ναι, βεβαίω είναι πρόκληση, που, αυτό που λέτε είναι πρόκληση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Αυτό δηλαδή σε σχέση με τη διασύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Αλλά θα πρέπει να, έχουμε ανάπτυξη και να δούμε τι θα γίνει με τι θέσει εργασία. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να μην ε, έχει ανάπτυξη. Δηλαδή, τη στιγμή που υπάρχει τόσο ταχεία ανάπτυξη στην Ασία, σε άλλες περιοχές ε, του κόσμου, στην, ε, ε, στην Νότια Αμερική, στην Μέση Ανατολή, δεν είναι δυνατόν εμείς με έναν διαρκώς γυράσκοντα πληθυσμό να μην μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό είναι βεβαίως η επένδυση σε δεξιότητες. Και είπα στην αρχική μου παρέμβαση ότι χρειάζονται κατά αυτή την έννοια πολύ περισσότερες επενδύσεις. Και είπα επίσης ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, την πρόορια εγκατάλειψη του σχολείου και των σπουδών. οι άνθρωποι φεύγουν από την αγορά εργασίας γιατί γερνούν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν όμω άνθρωποι οι οποίοι είτε φεύγουν από την αγορά εργασία είτε απλούστατα δεν μπαίνουν καν στην αγορά εργασία γιατί δεν έχουν αρκετέ ικανότητε, δεξιότητε, γνώσει. Επομένως, η στρατηγική ε, του 2020 ε, θα ε, έχει επιτυχία μονάχα εάν ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι πρέπει να γίνει. Ε, για τη στρατηγική της Λισαβόνας είχαμε συμφωνήσει επί πολλών θετικών στοιχείων. Τώρα, τώρα, εάν εσείς καταφέρετε να πείσετε το Συμβούλιο ότι χρειάζεται πιο αποτελεσματικό benchmarking στα πράγματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως δεν μπορώ να το πω εγώ. Όμως είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε πιο δεσμευτικές στρατηγικές και από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι εμείς επαφιέμεθα στα κράτη-μέλη. Είναι δικές τους αρμοδιότητες επίσης τα, τα, τα ζητήματα του, της ε, διαβίου μάθησης, εκπαίδευσης ε, κτλ. Και ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξω. Είναι για να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Λίν. Ε, ποιος θα πληρώσει την ε, ενσωμάτωση και πώς θα την κάνουμε. Έχουμε μια, ένα σχέδιο συμφωνίας το οποίο έχει υποβληθεί στα μέλη μας ε, προς έγκριση. Βεβαίως δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τις ε, ε, επιχειρήσεις ή τον κόσμο. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πείσουμε, ε, να ευαισθητοποιήσουμε τους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε με τη σειρά τους να κινητοποιηθούν για να λύσουν τα προβλήματα. Συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, και συνδικάτων. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Βεβαίως δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε και να αναγκάσουμε ε, ανθρώπους ε, οι επιχειρήσεις, αλλά μέσω μιας καλής συνεργασίας νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπενασί. Allora, per cercare di stare nei minuti parlo italiano. Αφού έχω μόνο τέσσερα λεπτά, νομίζω ότι θα μιλήσω ιταλικά, θα πάει πολύ πιο γρήγορα. <laughs> και βοήθειά μα λένε οι διερμηνείς. Ε, εν πάση περιπτώσει όλο αυτό με έκανε να χάσω και 25 δεύτερα. Θα πάω ακόμα πιο γρήγορα. Λοιπόν, Λοιπόν, δεν μπορώ να καταφέρω να αντιδράσω ε, στις ερωτήσεις που άκουσα με τη σειρά. Ε, θα προσπαθήσω όμως όσο γίνεται πιο γρήγορα να το κάνω. Σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, θα πω ξεκινώ από αυτά που είπε η Πρόεδρος θα πρέπει να δούμε σε αυτά τα τρία σημεία με μεγαλύτερη μάχη για τη νέα αυτή διακυβέρνηση διαχείριση και που επιτυγχάνει να περάσει αυτό το σχέδιο. Να δούμε και το επίπεδο αυτής της διαχείρισης. Έχουμε στοιχεία σε τελευταία δύο χρόνια, σε περίοδο κρίσης, τρομερά για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ορισμένες περιφέρειες και Δήμους. Όσο μικρότερη επιχείρηση, τόσο σε τοπικότερο επίπεδο είναι. Και σε περιφέρειες που είχαμε ένα κοινωνικό διάλογο, μια παρόμοια διαχείριση, πώς το πω τώρα, μια επικουρικότητα πραγματικά προωθημένη σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι το σημαντικό για τις ό,τι θέλετε, όσε συνεδριάσεις μπορούμε να οργανώσουμε, αλλά επί επιτόπου εκεί δεν θα πετύχουν τίποτα θετικό και θα υπάρξει ένα σχέδιο. Και αυτός που προωθεί το σχέδιο είναι το 1% οι επιχειρήσεις, να μην σας πω το 100%. Έτσι, ε, ίσως νομίζετε ότι είναι μεροληπτό. Τέλος πάντων, ε, από το 99 μπορώ να πεταχτώ στο 100. Εδώ αυτό έχει κατά γενικές γραμμές. Για να δούμε τώρα ειδικότερα τι γίνεται. Πώς θα τα καταφέρουμε και λέω στην Επιτροπή να ξεκινήσει ένα παρόμοιο πολύ σημαντικό σχέδιο. Λίγο πριν από την κρίση δεν είναι και τόσο τυχερή. το think, το think small first. Αυτό θα πρέπει να έχουμε, δηλαδή τα μικρά σχέδια και μετά να εφαρμοστούν σε κάθε επίπεδο. Έτσι, πρώτο και δεύτερο σημείο, αυτά συνδέονται άμεσα. Πάνω σε αυτά, ε, να πρέπει να σκεφτούμε πρώτα τα μικρά-μικρά, να μην είναι έτσι μεγάλα λόγια, φραστικά πυροτεχνήματα και φλιαρίες. Μια εφαρμογή των πολιτικών να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητα να αναπτυχθούν, έτσι. Και μετά άλλα σημεία για να δούμε τώρα την ανάπτυξη και της, ε, την αύξηση της απασχόλησης. Και τρίτο σημείο για καλύτερη εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών ε, μέχρι σε ιδιαίτερα τοπικό επίπεδο και αναφέρομαι στην Επιτροπή και πάλι. Έχουμε να δούμε τι ε, πώς επηρεάζουν τα πράγματα όλη η οργάνωση και θα απασχολήσει και τον Επίτροπο Μπαρνιέ ε, για αυτή την κοινωνική ρύθμιση διευθέτηση. Εδώ λοιπόν για αυτό τον αντίκτυπο λοιπόν. Θα πρέπει να δούμε αυτή την ανάλυση, όλα αυτά που είναι πίσω από ότι εδώ μελετάμε στις Βρυξέλλες και όχι μετά για να δικαιολογήσουμε για το τι έγινε. Αν αυτά τα πράγματα, αυτά τα τρία σημεία μπορούν να εφαρμοστούν, τότε θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ο χώρο τουλάχιστον κατά την απόψή μου, στι μικρές επιχειρήσεις, εκείνες που προωθούν καινοτομίε μπορούν να αναπτυχθούν, να μεγαλώσουν και πρόκειται ε, για ένα χώρο που υπάρχουν συνεχεί αλλαγέ, βελτιώσει κλπ. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα παραδείγματα θέματα, ένα όμως μόνο που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, λέμε τώρα ότι καθιστούν έτσι πληρωμές και όλα αυτά δείχνονται αναποτελεσματικά ενώ έχουμε καθυστερήσει δυόμιση χρόνια. Ή μιλάμε για ένα σχέδιο από τη στιγμή που τα μέσα, τα εργαλεία δεν μας επιτρέπουν από την αρχή να το καταστήσουμε κάτω συγκεκριμένο. Πώς ακόμα 17, τι να σας πω τώρα. Ουφ, δεν καταφέρω να σας πω και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Οι κοινωνικές πολιτικές ε, με τις υπόλοιπες πώς θα συνδυαστούν. Εμείς ε, αγριέψαμε όταν είδαμε και το επαναλάβαμε ότι αυτό το ε, νέο 2020. Δεν μας πήγαινε γιατί δεν υπήρχαν εμπορικές κοινωνικές πολιτικές. Θα μπορούσαμε να ε, απτύξουμε αυτό ιδιαίτερα για την Ινδία και την Κίνα. Αλλά εδώ, εδώ ξέρεις, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τα επόμενα 10 χρόνια και να δώσουμε 7 εβδομάδες, εντάξει, είναι προσπάθεια 8 τέλος πάντων. Ε, γιατί μπήκαν στη μέση και διακοπέ των ε, Χριστουγέννων για μια σοβαρή απάντηση. Θα κάνουμε τώρα, θα, μιλάμε μόνο θα, και τίποτα άλλο. Και εμεί αγριέψαμε και είπαμε θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ακούστε, <laughs> ναι, ναι, δώσε τη μάχη σας σήμερα το απόγευμα. Ραφ, ο κύριος Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Θα μπορούσα να μιλήσω γερμανικά. To finish in Italian. So, first... Αλλά θα σας καθυστερήσω, μάλλον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς που με ενισχύσατε όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες. Τόνισα την ε, μεγάλη σημασία τους και χαίρομαι που τα αναγνωρίζετε, διότι σε περίοδους κρίσεων αυξάνεται η σημασία τους περαιτέρω. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, στις περισσότερες ερωτήσεις. Καταρχάς, τι θεμελιώδη προέγγιση. Εάν θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό το έγγραφο ή να το ρίξουμε στα σκουπίδια. Ε, είναι δύσκολο να απαντήσουμε με ένα ναι ή ένα όχι. Όπως είπες και ο Ανδρέα, είναι πολύ δύσκολο να συγκεράσουμε τη στρατηγική όλων των επομένων δέκα ετών ε, χωρίς ορισμένες γενικότητες. Πρέπει λοιπόν να... Ε, είναι ευέλικτη η απάντησή μας, διότι πολλά θέματα δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τουλάχιστον από πλευρά CEEB θα πρέπει να διαγράψουμε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική ε, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε έναν ε, ε, επικοδομητικό διάλογο για τη στρατηγική του 2020. Όσον αφορά τώρα τα εργαλεία, τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, εδώ θα μπορούμε να χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσουμε ε, γενικά μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση, διότι αν εγώ παρουσίαζα μια τέτοια γενικόλογη έκθεση στη Γενική Συντέλευση του οργανισμού μου, δεν θα περνούσε, μάλλον θα με διώχνανε. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, όσον αφορά την απασχόληση να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ε, λίγες δεξιότητες, που έχουν λίγες ικανότητες ή προσόντα και να μπορέσουμε να τους προωθήσουμε. Για την οδηγία του χρόνου εργασίας που αναφέρθηκε θα ήθελα να συμφωνήσουμε σε μία συζήτηση αναθεώρησης αλλά δεν ξέρω ακόμα σε ποιο επίπεδο θα γίνει αυτή η διαβούλευση για την αναθεώρηση. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα σε τι επίπεδο πρέπει να γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Και βεβαίω, αν γίνει αναθεώρηση αυτή τη οδηγία, πρέπει να γίνει σε διατομεακό επίπεδο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για την οργάνωσή μου, για το ΣΥΠ, ήταν η συζήτηση του άρθρου 14 της συνθήκης ε, για τις δημόσιες υπηρεσίες και πάλι και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο συνεδρίασε για πρώτη φορά η Ειδική Επιτροπή Δημοσίων Υπηρεσιών ορισμένα από τα μέλη ήταν παρόντα μάλιστα και παρουσιάσαμε την εμπειρική εικόνα των δημοσίων υπηρεσιών σήμερα, αλλά η εμπεριστατωμένη έκθεσή μας, όπως είπα, θα παρουσιαστεί το Μάρτιο. Πρέπει λοιπόν το Μάρτιο να παρουσιάσουμε το μέλλον των δημοσίων υπηρεσιών, διότι νομικά ή νομοθετικά μέτρα δεν οδηγούν αυτόματα σε λύσεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια και οικονομική ασφάλεια. Λοιπόν, πρέπει να είναι εξασφαλισμένες οι δημόσιες ε, υπηρεσίες και από απόψεις χρηματοδότησης και από απόψεις νομικής για να μπορέσουν να παραμείνουν ε, επικοδομητικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ορισμένες ερωτήσεις ε, απευθύνθηκαν σε μένα και θα τις απαντήσω. Η οδηγία για τις ώρες εργασίας. Λέει ο κύριος Μόγκς. Ε, πιστεύω ότι έχει συζητηθεί πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για την ε, υποστήριξή του. Έχει συζητηθεί η οδηγία αυτή και στο Συμβούλιο Υπουργών πολλές φορές. Υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή και σε ορισμένα στελέχη της Κομισιόν ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να ε, καλύψουν το θέμα αυτό της οδηγίας. Δεν το πιστεύω, δεν συμφωνώ και ούτε προσφέρω την εθελοντική μου εργασία. Δεν είμαι εθελοντής της αναθεώρησης. Δεν πιστεύω ότι το θέμα αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων να το λύσουν αυτοί βλέπουμε ότι μεταξύ των κοινωνικών εταίρων υπάρχει μία σύγκληση απόψεων και η Business Europe έχει επισημάνει ότι υπάρχουν συνήθως προβλήματα εφαρμογής, όχι προβλήματα προσέγγισης. Μην Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και το έχουμε συζητήσει βεβαίως και με ενώσεις εργοδοτών. Ε, και εάν θέλουμε να είμαστε για το 2020, ρωτώ, θα έχουμε θεσμικές αλλαγές την επόμενη δεκαετία. Η απάντηση είναι βέβαιη. Οι κρίσεις, τέτοιες μεγάλες κρίσεις, ε, οικονομικές κρίσεις, οδηγούν συνήθως σε ριζικές αλλαγές. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, αν θα βρεθεί κάτι καινοφανές, θα προκύψουν καινούργια θεσμικά όργανα ή θεσμικά πλαίσια. Δεν το πιστεύω. Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορούμε ε, να βελτιώσουμε οπωσδήποτε το διάλογο, την επικοινωνία μας. Το είπα και στον κύριο Τρισέρ ε, της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας ότι υπάρχει έλλειμμα στην κοινωνική, στη στρατηγική της κοινωνικής πολιτικής και συμφώνησε μαζί μου. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές. Και η βασική ερώτηση στο μυαλό μου είναι γιατί αυτό το 2020, πώς ας πούμε επιλέξαμε αυτή τη δεκαετία, τι, τι θέλουμε να επιδιώξουμε γιατί όλος αυτός ο χαλασμός. Η Λισαβόνα έχει σαφείς στόχους και διατάξεις και είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας στη στρατηγική της Λισαβόνας. Είχε ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό, στις διάφορες στρατηγικές κλπ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτός ο χαλασμός για το 2020 και αυτή τη στρατηγική. Το ερώτημα το ουσιαστικό είναι τι επιδιώκουμε με αυτή την άσκηση στρατηγικής 2020. Ας πούμε τουλάχιστον ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε την γενική εικόνα της μελλοντικής Ευρώπης όσον αφορά την πορεία της στη βιομηχανία, την πορεία της στο να γίνει πιο πράσινη και ένα γενικό όραμα. Αυτό είναι, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε γενικά σε ένα όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, ε, το καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ε, τέσσερις ε, ομιλητές. Πρόκειται για συζήτηση η οποία βεβαίω τώρα ξεκινάει. Φτάνουμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της πολιτικής, της, των εργασιών μας ε, και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία ε, Σεν Τζόουν. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής απασχόλησης. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την δυνατότητα να μιλήσω εδώ σε εσά. Λέγομαι Σιαν Τζόουνς και είμαι συντονίστρια στρατηγικής της EAPN. Ε να σας πω ε, ποια είναι η κοινωνική πλατφόρμα. Είμαστε η μεγαλύτερη ένωση κοινωνίας των πολιτών ε, που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την κοινωνική ε, αδικία και να προαγάγουμε την συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρώπη. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο 42 πανευρωπαϊκών δικτύων μη κυβερνητικών οργανώσεων και προσπαθούμε να αναπτύξουμε την εταιρική σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις έτσι ώστε ε, να προωθήσουμε την ε, ε, βελτίωση της ζωής και τη μεγαλύτερη ελληνική. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο ε, στη διάθεσή μου και επομένως ε, πρέπει να σας πω ότι από τη στιγμή που μιλάμε για τη στρατηγική 2020, να σας πω ότι το κυριότερο μέλημά μας είναι η ερώτηση, μα τι είναι αυτή η στρατηγική. Ε, εμείς βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι είναι μια φιλόδοξη στρατηγική και καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή πρόκειται για μια στρατηγική η οποία προτίθεται να βάλει στο κέντρο των στόχων και των προγραμμάτων την κοινωνική ε, την ενδυνάμωση, την ακύρωση του κοινωνικού αποκλεισμού και τα κοινωνικά ζητήματα γενικότερα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει ε, πολύ ικανοποιητικά βήματα. Δηλαδή τα ε, έγγραφα τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα είναι γρήγορα, είναι μάλλον κακογραμμένα ε, και εν πάση περιπτώσει στην ουσία αυτό που διαπιστώνομαι είναι ότι δεν έχει ανασχεθεί ακόμα η πορεία του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη και τα προβλήματα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Επίσης διαπιστώνομαι ότι η διαδικασία διαβούλευσης δεν είναι η πλέον προσήκουσα, δεν είναι σωστή δεν μας ε, ικανοποιεί και τα διαβουλευτικά έγγραφα ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, απασχολήσουν σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην ουσία πρόκειται για μια αδιαφανή και μη δημοκρατική διαδικασία και μιλάμε προς Θεού εδώ για την κατάσταση η οποία, για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για τα επόμενα δέκα χρόνια και θα ισχύσουν για τα επόμενα δέκα χρόνια. Κατά την άποψή μας υπάρχει ένα σαφές ερώτημα σχετικά με την διασύνδεση ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μέχρι τώρα αυτή η διασύνδεση είχε θετικό πρόσημο ή όχι. Κατά την άποψή μας η ανάπτυξη δεν οδηγεί αυτόματα ε, σε ε, θέσεις εργασίας. Βεβαίως δεν οδηγεί ε, μαθηματικά και σε μείωση των θέσεων εργασίας ή μεγαλύτερο κοινωνικό αποκλεισμό. Το, το ζήτημα είναι να δούμε ε, με ποιο τρόπο μπορούμε να διασυνδέσουμε την ανάπτυξη με, τη θέση εργασία, με τις θέσεις εργασίας, γιατί δεν υπάρχει αυτοματισμός ε, στην ε, σχέση αυτή. Επομένω, αυτό που ρωτάμε εμεί είναι μάθαμε το μάθημά μα, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε την αίσθηση ότι μάθαμε το μάθημά μα από το παρελθόν. Κοινωνική συνοχή, ε, η κοινωνική συνοχή, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, ε, τα βλέπουμε μάλλον σαν εργαλεία, ενώ ε, πρόκειται για ρήτρε, οι οποίε ήδη υπάρχουν στη συνθήκη τη Λισαβόνα και οι οποίε δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Επίσης μας απασχολεί και η υπερβολική έμφαση που δίνεται εις την απασχόληση ως πανάκια, ως λύση για τα πάντα. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και οι οποίοι παρόλα αυτά ε, είναι φτωχοί. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται εκτός των ε, όρων ε, απασχολησιμότητας και επομένως δεν μπορούν να μπουν στην αγορά εργασία. Αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί μονάχα η εργασία, γιατί μονάχα η απασχόληση, τι γίνεται με τους νέους, τι γίνεται με τους ηλικιωμένους, τι γίνεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τι γίνεται με τον, με τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό. Υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα τα οποία δεν αναφέρονται καθόλου. Πολλά ωραία λόγια ακούμε. Πολλά ωραία λόγια ακούμε και για την governance, για τη διακυβέρνηση, αλλά επί του δεν δεν βλέπουμε τίποτα συγκεκριμένο. Πώς θα αναμειχθεί, σοβαρά εννοώ να αναμειχθεί το Κοινοβούλιο ε, με την διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ε, κοινωτικό. Ποιες είναι οι προτάσεις μας τώρα. Πρώτα απ' όλα εμείς έχουμε ε, πέντε μαθήματα τα οποία θα πρέπει να ε, ε, μάθουμε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια κοινωνικά υφόρο στρατηγική. Πολλά ωραία λόγια έχουμε ακούσει και για αυτό το θέμα, αλλά σχεδόν τίποτα δεν έχει γίνει που να ξεπερνάει λίγο τα εσκαμένα. Δεύτερον, λέμε ότι θα πρέπει να πάμε πέρα από τις θέσεις απασχόλησης σαν μοναδική κοινωνική απάντηση να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την ένδια και, την, και τον αποκλεισμό. Ε, θέλουμε να ενδυναμωθεί το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Ε, θέλουμε ε, να διασφαλιστεί ένα σωστό επίπεδο αμοιβή και εσόδων. με ελάχιστο εισόδημα για αξιοπρεπή εργασία. Ε, πρόσβαση σε ασφαλή εργασία και πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες οι οποίοι και από την αρχή έχουν αναγνωριστεί σαν πυλώνες για, τον, ε, για, για την κοινωνική ολοκλήρωση. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε ποιοτικέ θέσεις εργασίας και μια ευρωπαϊκή στρατηγική η οποία αυτογενώς να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας βλέπουμε ε, στην προσέγγιση της ε, στρατηγικής 2020 ότι ε, το κύριο όχημα είναι η οικονομία, η αγορά. Βλέπουμε μια στρατηγική η οποία είναι σαφώς οικονομικά προσανατολισμένη. Θα ήθελα τώρα να μπω σε λεπτομερία σε κάποιες από τις προτάσεις. Αυτό που προτείνουμε εμείς ε, σαν οικονομική στρατηγική είναι οι άνθρωποι πρώτα. Βεβαίως θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, βεβαίως λέμε ότι η οικονομία ε, είναι ένα εργαλείο ε, το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε απέναντί μας που είναι η φτώχεια. Αλλά λέμε ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν συνολικά οι ανισορροπίες και οι ανισότητες. Πού όμως βρίσκονται τα στοιχεία για το ξεπέρασμα αυτών των προβλημάτων μέσα στη στρατηγική. Δεν τα βρίσκουμε, δεν τα βλέπουμε. Επίσης, όσον αφορά το περιβάλλον, ε, έχουμε πέντε ε, αρχές ε, οι οποίες τίνουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αηφόρα ανάπτυξη, στην δημοκρατία, η οποία θα καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του περιβάλλοντος και στην ανάληψη συνολικής ευθύνης. Όσον αφορά τώρα τις εργασίες, είπαμε ότι θα πρέπει να πάμε πέρα από την απασχόληση σαν την μοναδική κοινωνική απάντηση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι νέες στρατηγικές προτεραιότητες, γιατί η μέχρι τώρα οι στόχοι μας δεν είναι ε, σωστοί. Λέμε ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε την, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις ανισότητες, αλλά βεβαίως χρειάζεται και ε, κοινωνική ε, συνένεση αλλά και κοινωνικός συντονισμός που θα αποτελέσει κεντρικό σημείο. Επίσης, χρειαζόμαστε ισχυρά κοινωνικά δικαιώματα σύμφωνα με το ε, Ευρωβαρόμετρο 64% των Ευρωπαίων λένε ότι θέλουν καλύτερη ε, κοινωνική Ευρώπη οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε μια οδηγία όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα και τη διασφάλιση αυτού του ελαχίστου εισοδήματος. Επίσης ε, θα πρέπει να ε, ε, υπάρχει διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέλος, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, συμμετοχή στην, της κοινωνίας των πολιτών το Κοινοβούλιο πιστεύω ότι είναι η καλύτερη, το, το, ο καλύτερος θεσμός ε, που μπορεί να προωθήσει πραγματικά, να πιέσει προς τη σωστή κατεύθυνση τους κοινωνικούς εταίρους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την παρουσίαση αυτή και έτσι ακούσαμε τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Ξεκινάει η συζήτηση. Εντάξει, δεν θα λάβουν ε, όλοι το λόγο, αλλά κάποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να παρέμβουν. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Κύριος Κλάρκ ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω το, το, τον ελάχιστο μισθό, την ελάχιστη αποζημίωση και μια ευρωπαϊκή οδηγία σε αυτό το θέμα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυτή τη ρύθμιση και η χώρα μου, το Ενωμένο Βασίλειο, για το, την ελάχιστη υποζημίωση. Όμως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε μία απόφαση που έλεγε ότι σε τέσσερις χώρες εργοδότες μπορούσαν να πληρώσουν λιγότερο από το ελάχιστο ποσό τους εργαζόμενούς τους και έτσι κατέστρεψαν την κοινή αντίληψη και την σύγκληση των απόψεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίντ μετά η κυρία Σρέντερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για την... Σας ευχαριστώ ε, κυρία Τζόνς για την έξοχη παρουσίασή σας. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα με αυτό το έγγραφο για τη στρατηγική 2020 ε, έχει πάρα πολλά ελλείμματα, πάρα πολλά θέματα δεν καλύπτονται. Ε, ε, σημαντικοί τομείς έχουν παραληφθεί και γενικά δεν αναφέρει συγκεκριμένα μέτρα της στρατηγικής αυτής. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση, αυτό το έγγραφο 2020 είναι αποτέλεσμα μιας αντίληψης ότι κάτι πρέπει να φτιάξουμε, κάτι πρέπει να παρουσιάσουμε και να δημοσιεύσουμε και έτσι στα γόνατα έγινε αυτή η έκθεση που βλήθηκε αυτό το έγγραφο άκουσα από πολλούς ότι δεν υπήρχε αναγκαίος χρόνος συζήτησης και διαβούλευσης για το τι πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε. Εάν θέλουμε τα επόμενα δέκα χρόνια να συνεχίσουμε ρεαλιστικά ή να διαμορφώσουμε ρεαλιστικές πολιτικές ε, πρέπει να ξανακάτσουμε και να μελετήσουμε τι θέλουμε. Ε, πιστεύω ότι αυτή η γρήγορη στο γόνατο μελέτη που έγινε δεν θα μας ωφελήσει καθόλου στο να επιλέξουμε συγκεκριμένα μέτρα για τα επόμενα δέκα χρόνια δεν νομίζω ότι το έγγραφο αυτό είναι επαρκές. Στην πραγματικότητα είναι ανεπαρκέστατο και πιστεύω ότι η Κομισιόν πρέπει να το αναθεωρήσει και να προβάλλει συγκεκριμένες απόψεις. Η κυρία Σρέντερ, ευχαριστώ. Πολύ σημαντική παρουσίαση ήταν αυτή της ε, κυρίας Λίν διότι λείπει αυτή η πτυχή στην στρατηγική του 2020. Και δεν λείπει μόνο σε αυτό το έγγραφο που ανέφερα, αλλά και σε πολλά άλλα στρατηγικά έγγραφα στο πλαίσιο της Λισαβόνας. Ακούσαμε σήμερα ότι η προώθηση της κοινωνικής ε, ε, ενσωμάτωσης πρέπει να αποτελέσει ένα πρωταρχικό στόχο και η καταπολέμηση βεβαίως της, του κοινωνικού αποκλεισμού. Ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν καλύπτονται από καμία στατιστική ε, διότι δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα ή σε έναν ορισμένο τομέα. Άρα λοιπόν διαφεύγουν από τα στατιστικά μας στοιχεία και έτσι αποκλείονται κοινωνικά. Έχουμε λοιπόν στοιχεία τα οποία δεν είναι ακριβή και δεν ε, καλύπτουν πολλά άτομα, πολλούς πολίτες που βρίσκονται εκτός των γεγονότων και εκτός οποιασδήποτε στρατηγικής. Χαίρομαι λοιπόν που αναφέρθηκε αυτό το θέμα και ε, χαίρομαι που είπατε ότι αυτός ο αριθμός των κοινωνικών αποκλεισμένων, κοινωνικώς αποκλεισμένων πρέπει να βελτιωθεί, ε, πρέπει να μειωθεί το, το, ποσοστό αυτό βεβαίως και συμφωνώ απόλυτα. Επίσης είπατε ότι χρειάζονται νέες κατευθυντήριες γραμμές για μια δραστήρια πολιτική κοινωνικής ενσωμάτωσης όταν λέμε κατευθυντήριε γραμμές, ε, είναι πολύ γενικά μέτρα αυτά. Εδώ θα ήθελα πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Και τρίτον, τι προτάσεις έχετε για συγκεκριμένα ε, συγκριτικά στοιχεία, για το συγκεκριμένο benchmarking της στρατηγικής 2020. Ευχαριστούμε. Τόμας Μαν, πρώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εδώ μιλούμε μία διαφορετική γλώσσα από ό,τι φαίνεται. Ίσως η πρώτη στρατηγική της Λισαβόνας ήταν τόσο δύσκολη και τόσο υπερβολικά φιλόδοξη που δηλαδή θέλαμε να συγκριθούμε με τους Αμερικανούς που τελικά οπισθοχωρήσαμε και είπαμε ας επανέλθουμε στις ρίζες μας, ας επανέλθουμε σε αυτά που ξέρουμε. Ε, τώρα λοιπόν μιλάμε μία γλώσσα την οποία μπορούμε να, να καταλάβουμε και γι' αυτό εφαρμόσαμε μία πιο επιφυλακτική φωνή. Υιοθετήσαμε λοιπόν μία πιο κουρασμένη αν θέλετε προσέγγιση. Πολλές φορές ε, μας κατηγορούν ότι η οι ιδέες μας ε, δεν πέρασαν, δεν έφτασαν στους κατάλληλους αποδέκτες. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν γνωρίζετε ποιοι είναι αποδέκτες των ιδεών σας και αν γνωρίζετε εάν το ευρύ κοινό τις δέχεται ή τις απορρίπτει. Ο διάλογος που έχουμε με την κοινωνία των πολιτών. Εδώ χρειάζεται ένα εκατομμύριο υπογραφές για να ανεληφθεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι ποσοστά πρέπει να υιοθετήσουμε για να ε, μπορέσουμε να προωθήσουμε ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες. Έχουμε πει ένα εκατομμύριο. Όμως, ε, στη συγκεκριμένη εφαρμογή αυτού του μέτρου, αυτοί οι αριθμοί δεν συμπληρώνονται. Άλλο θέμα είναι η παγκόσμια ευθύνη. Ε, το global responsibility, αυτή η ευθύνη ε, και οι επιχειρήσεις συμμετέχουν βεβαίως σε, αυτό, διαμορφώνουν τη γενική εικόνα μας προς τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την παγκόσμια πραγματικότητα και δεν θα πρέπει να μας κατηγορήσουν ότι ζούμε σε απλησίαστες σφαίρες πολιτικής. Πάντοτε να είμαστε ρεαλιστές. Ευχαριστώ για τη θαυμάσια αυτή παρουσίαση της κοινωνικής πλατφόρμας. Έχουμε τώρα 20 χρόνια εμπειρίας στη συζήτηση πολλών μηχανισμών, μέτρων, πλαισίων, φορέων και τα λοιπά για τη αντιμετώπιση της φτώχειας. Και όμως είναι πολύ απογοητευτικό να βλέπουμε την ίδια παραδοσιακή προσέγγιση της Κομισιόν. Καταρχάς, η Κομισιόν φαίνεται ότι δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα νέα κριτήρια που έχουν ε, παγιωθεί πλέον στις συνθήκες ε, και στη συνθήκη της Λισαβόνας εδώ υπάρχουν οριζόντιες ρήτρε που έχουν συμπεριληφθεί με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων σε όλες τις πολιτικές. Δεν έχουμε λοιπόν αποδείξεις ότι η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη αυτές τις οριζόντιες ρήτρε. Σχετικά τώρα με τον Γενικό Συντονισμό της ανοιχτής μεθόδου, το μεγάλο πρόβλημα, και το έχω πει επανειλημμένως, είναι ότι αυτή η ανοιχτή μέθοδος δεν είναι διόλου ανοιχτή. Πρέπει να κάνουμε μία δημόσια συζήτηση για το τι προτείνεται και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Αυτή η έλλειψη πρόσβαση, ανοιχτής πρόσβασης έχει πολλές φορές ε, οδηγήσει την Κομισιό να αποτύχει στην επίτευξη των στόχων της δεν υπάρχει πίεση από τους ομολόγους μας. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε αναθεώρηση, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε, να ανοίξουμε ε, τις ε, πόρτες μας στο δημόσιο ε, έλεγχο, όχι στο δημόσιο έλεγχο, στο κοινό. Να ανοίξουμε τις πύλες μας, να, να, να ελευθερώσουμε την πρόσβαση έτσι ώστε να είμαστε ανοιχτοί προς τους πολίτες μας κυρία Σεντζόνς. Ευχαριστούμε που σε, που πέντε λεπτά, σε τέσσερα λεπτά θα απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, τις πέντε. Ευχαριστώ για τα ενδιαφέροντα αυτά ερωτήματα και παρατηρήσεις, θα απαντήσω σύντομα. Όταν μιλάω για ελάχιστο εισόδημα, μίλησα για ελάχιστο εισόδημα, όχι ελάχιστο μισθό. Εμείς ζητούμε στα πλαίσια της κοινωνικής ενίσχυσης ελάχιστο εισόδημα. Η σύστασή μας τώρα έχει συζητηθεί από το Συμβούλιο, το Συμβούλιο και, και η Κομισιόν έχει επιβεβαιώσει ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα ενός μήνυμου μισοδήματο για μια ξεπρεπή ζωή. Αυτή η αρχή, αυτή η βασική αρχή είναι θεμελιώδης για την αντιπεσόψη της κρίσης και αποτελεί μία πλατφόρμα για την εξέλιξη της ζωής του καθενός. Έχουμε και την νομική βάση να το εφαρμόσουμε. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι την βούληση των κρατών μελών ε, ε, για την εφαρμογή. Τώρα, τι περιθώριο έχουμε βελτίωσης ε, για την επίτευξη των στόχων. Εμείς θέλουμε τώρα ε, να παρουσιάσουμε τους συγκεκριμένους στόχους για την μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και της ε, ανισότητας. Η ανισότητα είναι μια μεγάλη πρόκληση και πολλές φορές δεν συζητιέται. Όμως η ανισότητα βλάπτει την κοινωνική συνοχή. Ε, φτώχεια λοιπόν κοινωνικός αποκλεισμός και ανισότητα. Το Συμβούλιο έθιξε το θέμα της ανισότητος, άρα λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης και γι' αυτό. Θα πρέπει στις ενσωματωμένες κατευθυντήριες γραμμές να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα έλεγα λοιπόν γιατί η βιασύνη ε, αυτής της στρατηγικής, ε, ε, γιατί τόσο γρήγορα να, περάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε χρόνο να τα σκεφτούμε λεπτομερώς και με μεγάλη προσοχή. Είχαμε πάρα πολύ θετική αντίδραση και θετικές εκθέσεις από τα κράτη-μέλη για την ε, εφαρμογή του συστήματος ελάχιστης αποζημίωσης, ελάχιστης αμοιβή ή μισθού. Ε, όμως σε άλλες περιπτώσεις το σύστημα δεν δούλεψε ικανοποιητικά. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε επαρκή χρόνο στη διάθεσή μας να συγκεράσουμε όλες τις απόψεις. Όσον αφορά τη συγκριτική μελέτη, το benchmarking είναι πολύ σημαντικό γιατί η Γαλλική Προεδρία έσπρωξε όλο αυτό το θέμα πέραν του ΑΕΠ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το ΑΕΠ για την ε, συγκριτική μέτρηση ε, της πρόοδου. Ε, χρειαζόμαστε καλύτερα περισσότερους παράγοντες περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, πέραν των οικονομικών, για να μελετήσουμε την πρόοδο, για να κάνουμε αυτό το benchmarking. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολλαπλούς αλλά και πολύμορφους δείκτες στοιχεία συγκρίσιμα για την φτώχεια τα έχουμε ήδη. Η πρόοδο λοιπόν μετράται όχι μόνο στα πλαίσια του ΑΕΠ, αλλά και όσον αφορά την ευημερία, τη μείωση της φτώχεια και την καταπολέμηση της ανισότητας. Η δουλειά έχει γίνει. Αυτό που χρειάζεται είναι η εφαρμογή. Και τέλος, ε, η παγκόσμια διάσταση είναι σημαντική και λείπει τελείως υπήρχε στις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά στο 2020, στη στρατηγική 2020 λείπει τελείως. Χρειαζόμαστε συνεκτικές πολιτικές, αλλά ε, πρέπει να, για να εφαρμόσουμε συνεκτικές πολιτικές πρέπει να μελετήσουμε και το ρόλο της ευρωπαϊκή Ένωσης παγκόσμια η παγκόσμια διάσταση λοιπόν έχει μεγάλη σημασία διότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις πιέζουν συνέχεια σε μια συνεκτική πολιτική, για μια συνεκτική πολιτική. Επίσης θέλουμε να αναφέρει η έκθεση αυτή το χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί ο συντονισμός των ανοιχτών μεθόδων μπορεί να λειτουργήσει σωστά, έχει λειτουργήσει σωστά. Ε, ίσως δεν λειτουργεί σωστά σε ορισμένα κράτη-μέλη, ε, αλλά όταν εννοούμε ανοιχτή μέθοδος, εννοούμε τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, όλων των stakeholders, και θα πρέπει ο συντονισμός αυτός ε, να βασίζεται σε πραγματικές ε, διαδικασίες, να συμπεριλαμβάνει και τη διάσταση των εθνικών κοινοβουλίων για να είναι επιτυχής. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα όσα συμπληρωματικά είπατε και μια κάποια στιγμή θα επανέλθουμε για να εκφράσουμε και πάλι τις σκέψεις μας και τις εργασίες μας ε, να, να διοργανώσουμε. Αυτά λοιπόν, ε, όπως σας είπα, δεν θα ασχοληθούμε με το 6 σημείο, θα πάμε στο σημείο 7, η συγγήτρια νομοδότησης, συντάκτη ανθρωπονομοδότησης, έχει το λόγο, κυρία γκράσλ που υπάρχουν πέντε γνωμοδοτήσεις απαλλαγής για τον προϋπολογισμό 2008. Ένα για την Επιτροπή και τέσσερα για άλλα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή μας. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτές τις γνωμοδοτήσεις. Η συγγητριά μας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γκρέσλεϊ. Γκρέσλεϊ λέγομαι. Εγώ προσπάθησα να πω ποια είναι αυτά τα ειδικά σημεία και της γερμανικής γλώσσας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να παρουσιάσω ορισμένα θέματα από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα αρχίσω με τη γνωμοδότηση για το ESF. Είναι τμήμα της έκθεσης Λιμπεράτσκι και αναφέρεται στα βασικά προβλήματα που έχουμε στη διαχείριση των διαθροτικών ταμείων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα τμήμα των διαθροτικών και έχει πολλά προβλήματα. Εγώ πιστεύω να ε, εγκρίνουμε, ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε μία απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, ορισμός των πληρωμών που έγινε χωρίς την απαραίτητη δικαιολόγηση είναι 11%. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες ε, ορισμένα θέματα τα οποία δεν είναι σωστά και ε, πιστεύω ότι η Επιτροπή αυτή ε, θα έκανε πάρα πολύ καλά εάν βγάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοταμείο από το από ολόκληρο το πακέτο των διαφορετικών ταμείων, διότι έχει συγκεκριμένε ιδιαιτερότητες ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αν θέλουμε να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, θα πρέπει η Επιτροπή μας να τονίσει τις ιδιαιτερότητες του Κοινωνικού Ταμείου. Θα πρέπει να απλωστεύσουμε και τους κανόνες και τους ελέγχους για να αποφύγουμε αυτές τις ατεσταλίες που σημειώνονται. Ε, πολλές φορές οι έλεγχοι αυτοί γίνονται από στελέχη τα οποία δεν έχουν καμία εμπειρία και δεν έχω την κατάλληλη εκπαίδευση. Ελπίζω να με υποστηρίξετε σε αυτή την πρόταση, διότι θέλω σαφώς να τονίσω την ιδιαιτερότητα αυτού του ταμείου. Μίλησα βεβαίως και με τη Γενική Διεύθυνση και με τον Επίτροπο. Εδώ και πέντε χρόνια είμαι μέλος της Επιτροπής Προεπιλογισμού και πιστεύω ότι έχει λίγο καταπιεστεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια των διαφορετικών ταμείων και αυτό είναι πάρα πολύ κρίμα. Θα πρέπει ε, να εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο έλεγχο των ευρωπαϊκών ε, πόρων, των πληρωμών και πιστεύω ότι και για την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα είναι πολύ καλύτερο να έχουμε συγκεκριμένες ε, ε, ε, εξηγήσεις για το πώς παρουσιάστηκαν αυτές οι ατασφαλίες. Η πολιτική μας λοιπόν πρέπει να είναι προληπτική, όχι διορθωτική εκ των υστέρων. Ώστε να μην χρειάζεται συνέχεια να καταφεύγουμε στην Όλαφ. Στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού έχουμε δει ότι μόνο 7% των υποθέσεων που χειρίζεται η Όλαφ ε, σε αυτές έχουν δοθεί συνέχεια. Ε, γι' αυτό λοιπόν ζητώ να διασφαλιστεί ότι οι υποθέσεις απάτης ε, θα παραπέμπονται σε εθνικές δικαστικές αρχές και έτσι θα ασκείται και δίωξη κατά των υπευθύνων. Αυτό θα βοηθήσει και πολύ στην ανύψωση της εικόνας της Ένωσης. Θέλετε να μιλήσω και για τα ευρωπαϊκά ιδρύματα, όλα μαζί, τα θέματα. Ωραία. Ευρωπαϊκό Ιδρύμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας. Αυτό είναι ένα θέμα και γενικά το Ευρωπαϊκό για την Ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, ασφάλειας και υγείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα βάσανο για την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ε, συνεχώς ε, συζητάμε για τα ιδρύματα αυτά, ε, μαζί, σαν ένα πακέτο. Γι' αυτό λοιπόν δύο από, τις, από τα τέσσερα αυτά, δύο από, τις, ε, από τα τέσσερα αυτά ιδρύματα ή κέντρα τα έχω επισκεφθεί και είναι μικρά σχετικά. Όμως ε, λειτουργούν βάσει πολύ διαφορετικού πλαισίου και έχουν προβλήματα με το καταστατικό τους. Δεν ξέρω καμία, κανένα ευρωπαϊκό ίδρυμα, οργανισμό ή κέντρο που να μην έχει προβλήματα ε, με το λογιστικό πλαίσιο και γι' αυτό συνεχώς υπάρχουν τριβές με το ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω μια επικοδομητική στάση και μια ενίσχυση του έργου των οργανισμών και των κέντρων αυτών που πολλές φορές ε, πνίγονται και δεν μπορούν να καταφέρουν ε, να ε, σεβαστούν τις αρμοδιότητές τους. Οι τέσσερις αυτοί οργανισμοί όλοι έχουν προβλήματα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα με το ETF που όσον αφορά τις προσλήψεις και θα παρουσιάσω μία δική μου τροπολογία για να μπορέσω να προβάλλω αυτό το πρόβλημα περισσότερο. Ορισμένα λαθάκια υπάρχουν συντακτικά τα οποία θα διορθώσω. Έχουμε λοιπόν, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με ένα κέντρο ή ένα ίδρυμα, αλλά έχουμε προβλήματα μέσου όρου, κατά μέσο όρο παρόμοιας φύσης και στους τέσσερις οργανισμούς ε, τα οποία αναφέρω στην έξεση μου. Θέλω τα προβλήματα που υπάρχουν να τα παρουσιάσω, διότι ε, αυτός είναι ο ρόλος μας, η εξέβρεση λύσεων. Σας ευχαριστούμε. Αυτές οι παρατηρήσεις για αυτά τα ιδρύματα για το προπολογισμό δεν ξέρω, ίσως άλλοι θα μπορούσαν να κάνουν παρόμοιες παρατηρήσεις, ορισμένες ενώσεις ή τοπικοί που πολύ συχνά παραπονιούνται εντάξει, για τη δυσκολία όλα αυτά να ισχύσουν για τους μικροφορείς. Ο Νταρντέν έχει δει στο λόγο και μετά για να δούμε ποιος άλλος συνάδελφος θα ήθελε. Λαμπέρ. Μάρκιν. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εισηγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι, τι παρατήρω σε αυτό το σχέδιο με αυτές τις νομοδοτήσεις που μας δίνει η συγγήτρια είναι λεπτομεριακές, ποιοτικέ, δείχνουν έτσι ποια είναι η άποψη του ηλεκτρικού συνεδρίου, αλλά θα ήθελα να κάνω παρατηρήσεις. Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τα προβλήματα, τα κενά και ότι θα πρέπει να δούμε ειδικότερα αυτό τον χαρακτήρα ε, τονίζονται στο σχέδιο εδώ και ακόμη όσοι επιτόπου εργάζονται μας ενημερώνουν ε, ότι η εκτέλεση αυτών των υποχρεώσεων σεβασμός ε, είναι και ένα δύσκολο έργο και χρειάζεται πολύ προσωπικό και να αφιερωθούν μέσα αυτά. Καλό θα ήταν δε να τονίσουμε ότι μερικές φορές είναι κάπως άκαμπτη όλη η διαδικασία ελέγχου. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε όταν μιλάμε για κυρώσεις. Το είπατε άλλωστε στην γνωμοδοτήσή σας για το κοινωνικό ταμείο αυτό είναι, αλλά για να δούμε τώρα και τα ιδρύματα. Να κάνω το εξή σχόλιο αφού διαβάζω τις απαντήσεις αυτών των ιδρυμάτων στις παρατηρήσεις του λεκτικού συνεδρίου, αλλά και όσα υπόθηκαν μετά από τη δημοσίευση του σχεδίου εκθεσής σας αποδεικνύουν ε, ότι υπάρχει διάθεση για την εκτέλεση του προπολογισμού και ότι σοβαρά λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Μην δώσουμε λοιπόν την εντύπωση ότι ε, είναι δακτυλοδεικτούμενα αυτά τα ιδρύματα από εμά. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι συμμορφώνται με τις συστάσεις ε, και όλα αυτά χρειάζεται να τα λάβουμε υπόψη μας στη γνωμοδότηση και στις πληροφορίες άλλωστε που μας προδίδονται και ίσως με μερικές τροπολογίες για αυτές δύο παραφηρήσεις για το κοινωνικό ταμείο για τα ιδρύματα αυτό να κάνουμε, αλλά σε επικοδομητικό πνεύμα να προσπαθήσουμε να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη μιας διαφάνειας και τον έλεγχο από την άλλη μεριά. Επίσης όμως για να μπορέσουμε να έχουμε πολιτική επιτόπου αποτελεσματική. Κύριε Λαμπέρτ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε βεβαίως την εισηγήτρια. στην γνωμοδότηση για το κοινωνικό ταμείο ε, ε, πολλά πράγματα βρίσκουν σύμφωνη, κυρίως και στην τελευταία παράγραφο όταν αναφέρεστε στην ε, ανάγκη ύπαρξης έκθεσης σχετικά με την απλούστευση της διαδικασίας. Νομίζω ότι πολύ συμφωνούμε. Είναι ένα καθολικό αίτημα. Υπάρχουν και, άλλα, και άλλοι προβληματισμοί, αλλά νομίζω ότι αυτοί θα απασχολήσουν ε, τον προϋπολογισμό. Πιστεύω ότι το πλαίσιο το οποίο έχετε ορίσει για, τις, ε, ε, για τους οργανισμούς είναι πραγματικά και τα ιδρύματα είναι πραγματικά σωστό και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι ζητούμε. διαπιστώνω ότι υπάρχει μία ε, ένταση ε, σε αυτά που λέτε και μας αφήνει να εννοήσουμε ότι είναι λίγο χειρότερη η κατάσταση και ε, θα υπάρξουν και κάποιες τροπολογίες οι οποίες ενδεχομένως θα εξισορροπήσουν λίγο αυτό το περιεχόμενο το οποίο είναι και πάρα πολύ αυστηρό πέρα από οποιουσδήποτε ε, κανόνες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι το περίπλοκο των ε, κανόνων. Σχετικά με αυτό το διαθεσμικό όργανο το οποίο θα επιβλέπει τα ιδρύματα, εκεί υπάρχουν ε, κάποιες επικρίσεις όσον αφορά τα καταστατικά και τους κανόνες βάσει των οποίων λειτουργούν τα ιδρύματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρκίν άλλος ε, ένας εισηγητής και τέλος. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την ε, εισηγήτρια για την πολύ σαφή περιγραφή της κατάστασης όσον αφορά πρώτα το κοινωνικό ταμείο. Μα ζητάτε να δούμε χωριστά ε, το κοινωνικό ταμείο, κυρίως διότι υπάρχουν καμιά φορά αποδέκτες οι οποίοι είναι πολύ μικροί και δεν θέλουμε να τους χάσουμε νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι αποθέκτες ε, του κοινωνικού ταμείου και ε, πού ακριβώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της υπερβολικής ε, γραφειοκρατίας. Από τη μία μεριά δηλαδή έχουμε τις, τους μικρούς που δεν καταφέρουν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα και από την άλλη μεριά ε, επιχαίους τίτλους εφημερίδων που φωνάζουν για απάτες ε, ε, όσον αφορά τα χρήματα αυτού του ταμείου. Επίσης αναφέρεται ότι η ΟΛΦΑ παρακολουθεί 7% των περιπτώσεων. Νομίζω ότι είναι απολύτως ουσιώδες γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πηχαίους τίτλους ε, εφημερίδων που αναφέρονται σε ε, απάτες ε, και αυτού του είδους οι διαδικασίες θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν και βεβαίως να δείχνουμε σε όλους ότι εμείς είμαστε απολύτως ανοιχτοί. Στο σημείο 6 αναφέρεστε σε αντιπαράθεση συμφερόντων ε, και αντικρουόμενα συμφέροντα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όσον αφορά τώρα τα ιδρύματα, είπατε ότι καμιά φορά είναι μικρά και επομένως δεν μπορούν πραγματικά να εκπληρώσουν τον ρόλο τους. Μ' αρέσουν αυτά που λέτε ε, για, το ίδρυμα, για τα ιδρύματα. Μ' αρέσουν οι προτάσεις που κάνετε έτσι ώστε να βοηθήσετε και τα ιδρύματα αυτά που δεν μπορούν να ε, τα βγάλουν πέρα και με τους προϋπολογισμούς και αυτά. Ε, βεβαίως ε, είναι γεγονός ότι καμιά φορά οι απαντήσεις που δίνουν σε διάφορες προκλήσεις τα ιδρύματα αυτά είναι έγκαιροι, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πλήρης και σωστή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άπιου τελευταία εγγεγραμμένη. Η κυρία Ράπτη τώρα. Η κυρία Ράπτη και μετά η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ε, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για τη δουλειά που κάνουν και να τους ευχηθώ καλή δύναμη για παρακάτω γιατί εδώ είναι η πρώτη κουβέντα που γίνεται. Ε, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για αυτά τα Ινστιτούτα, εγώ στο μυαλό μου έχω τους Ευρωπαίους πολίτες τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, τους Ευρωπαίους μαθητές, τους Ευρωπαίους καταναλωτές, τους Ευρωπαίους δάσκαλους. Ε, με άλλα λόγια, τα ιδρύματα αυτά έχουν δημιουργηθεί ώστε η δουλειά που κάνουν να φτάνει και να ωφελούνται από αυτήν τη δουλειά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό θέλω ε, να τα δούμε με συμπάθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε συγχωροχάρτη σε οτιδήποτε δεν είναι σωστό από τις ενέργειές τους. Όμως θέλω να τα δούμε με πραγματική συμπάθεια. Και νομίζω ότι το αξίζουν γιατί εγώ είδα, όπως φαντάζομαι όλοι μας, τις απαντήσεις που έχουν δώσει και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και το ETF στις ενστάσεις που αναφέρονται στην αρχική εισήγηση που έχει γίνει. Ε, αυτές εδώ τις απαντήσεις και τις πληροφορίες που έχουμε από τα ιδρύματα αυτά θα ήθελα, εάν γίνεται, να ληφθούν υπόψη στην τελική έκθεση. Και αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι τους οργανισμούς αυτούς, αυτά τα Ινστιτούτα πρέπει να τα βοηθήσουμε να κάνουν καλύτερη δουλειά, γιατί αυτή η δουλειά επιστρέφει σε μας. Ε, νομίζω ε, επίσης ότι καλύπτομαι, αισθάνομαι να καλύπτομαι από τις απαντήσεις που δίνουν και για το σημείο 5 της έκθεσης, ειδικά για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, είναι ένα ίδρυμα, θυμίζω, το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Προέρχομαι, είμαι ευρωβουλευτής που προέρχομαι από την Ελλάδα και έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, όπως επίσης νομίζω ότι υπάρχει καλή συνεργασία και με το μεταξύ του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και του ETF. Ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να είμαι έτσι ε, ξεκάθαρη ε, όσο μπορώ και εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις μέσα από τροπολογίες και με την πολιτική μου ομάδα να βοηθήσουμε ώστε οι οργανισμοί αυτοί να εργαστούν καλύτερα. Αλλά θα παρακαλούσα πολύ την εισηγήτρια να δείξει όλη την καλή της διάθεση και να είναι περισσότερο ανοιχτή σε αυτά τα ιδρύματα, γιατί αισθάνθηκα από την αρχική της τοποθέτηση μια απόσταση και ένα αυστηρό βλέμμα παραπάνω από αυτό που ίσως θα έπρεπε. Ευχαριστώ και εύχομαι καλή δουλειά για την συνέχεια. Σα ευχαριστούμε. Η συγγήτρια μήπω θα ήθελε να ολοκληρώσει με την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους. Ειλικρινά, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τις διαδικασίες ελέγχου σε αυτού τους οργανισμούς. Δεν είναι μόνο τέσσερι. Ε, έχουμε και άλλες τρεις ε, για το χρηματοπιστωτικό σύστημα πολλές, ε, λοιπόν, πολλά λοιπόν κέντρα ή οργανισμούς ή ιδρύματα ή Ινστιτούτα και σε, ορισμέν, σε μία από αυτές τις ε, οργανώσεις έχουμε μία υπέρβαση 4.500%. Ε, έχουμε λοιπόν σημαντικά προβλήματα ελέγχου και ατασταλιών. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι συμπαθητική και να απαντήσω με συμπαθητικό τρόπο. Ναι, βεβαίως πρέπει να ζήσουμε με αυτά τα κέντρα, με αυτούς τους οργανισμούς. Αυτή που λειτουργήσε θαυμάσια είναι ε, αυτή της, που, που είχε την έδρα της και στην Ελλάδα μάλιστα, η οποία λειτουργήσε εξαιρετικά ικανοποιητικά bitten, Θα πρέπει λοιπόν ε, να προχωρήσουμε μαλακά, ε, να μην, τους, να μην τις πνίξουμε ε, και να τις πάρουμε από το λαιμό. Πρέπει να δείξουμε, να ακολουθήσουμε μια συνετή και ήπια αλλά μεθοδική στάση. Δεν είμαι κατά των κέντρων ή των Ινστιτούτων αυτών. Γεγονός όμως είναι ότι η πραγματικότητα μας πιέζει να ρωτήσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ένα Ινστιτούτο 80 ή μάλλον στην ελεγκτική υπηρεσία 80-90 άνθρωποι και πρέπει να εκτελέσουν όλους αυτούς τους απαραίτητους ελέγχους. Καταρχάς λοιπόν πρέπει να έχουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία που χρειάζεται και απ' την άλλη πρέπει να βοηθήσουμε ε, τα ιδρύματα αυτά. Ε, προσπάθησα λοιπόν να καταγράψω τις ε, απόψεις των συμβούλων, των διευθυντικών στελεχών, του management δηλαδή, των κέντρων αυτών ε, και όλοι μου εξέφρασαν παράπονα για τις διαδικασίες ελέγχου. Όλες, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, αυτά τα Ινστιτούτα, στο τέλος του χρόνου έχουν περίσευμα χρημάτων. Αυτό που θέλω εγώ να επιδιώξω είναι να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα. Ε, τι νόημα έχει να τα να κάνουν αυτές τις οικονομίες, είτε είναι ηθελημένες είτε αθέλητες και μετά τον επόμενο χρόνο να μην μπορούν να ξοδέψουν αυτά τα λεφτά. Πρέπει λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα λογιστικά να δαπανίσουν τα χρήματα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους. Ε, και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες ε, επικρίσεις που εκφράστηκαν και πρέπει να δεχθούν την κριτική αυτή τα ιδρύματα αυτά. Κανένας δεν θέλει να σκοτώσει αυτά τα ιδρύματα. Όλοι θέλουμε να συνεχίσουν τη ζωή τους, και, αλλά να λειτουργούν σωστά και να ανταποκρίνονται στο στόχο τους. Εγώ είμαι στο πλευρό σας. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις, ε, τα ιδρύματα αυτά να μπορέσουν να σεβαστούν το πολύ περίπλοκο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο Υπάρχουν όμως κανόνες επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει. Άρα λοιπόν πρέπει αυτούς τους κανόνες να τους τηρούν. Ε, με παρακαλέστε να εκφράσω, να, να, να σχολιάσω την ε, διάσταση των συμφερόντων που υπάρχει, τη διαφορά αντιπαράθεση συμφερόντων ε, μεταξύ του στόχου των ιδρυμάτων αυτών και της διάθεσης των χρημάτων πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν εκφράζουμε ε, επικρίσεις. Εγώ δεν ε, διενεργώ τους ελέγχους και αν θέλουμε να κατηγορήσουμε για απάτη, ε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν τόσα επίπεδα ελέγχων και είναι και τέτοιο το κόστος του ελέγχου που πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά βήματα. Έχω συζητήσει και με τους τοπικούς φορείς που είναι αποδέκτες ε, κοινωνικών ε, πόρων και μου λένε ότι πολλές φορές ε, τα, τα κονδύλια αυτά δεν απορροφώνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, μη μου παρεξηγείτε, εγώ δεν έχω τίποτα κατά των ιδρυμάτων ή των κέντρων αυτών. Όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότιμη μεταχείριση και να ακολουθήσουμε ε, μία μετριοπαθητική, ε, μετριοπαθή συγγνώμη, τακτική. Λοιπόν, ισότιμη μεταχείριση όλων αυτών των κέντρων και ιδρυμάτων και ε, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την σωστή επιβίωσή τους. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Θα επανέλθουμε νομίζω και για τη διαχείριση όλων αυτών. Θα έλθουμε, θα είμαστε σε επαφή με τον εκπρόσωπό τους ε, αύριο από τις 3 το απόγευμα και μετά. Είναι γνωμοδοτήσεις αυτές ε, παρόμοιες και η Επιτροπή Αρμόδια Προϋπολογισμού θα ψηφίσει 22 Μαρτίου. Θα έχουμε το εξής διάγραμμα. Μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου τροπολογίες προς υποβολή. Υιοθέτησή τους. Ε, για να δούμε τι γίνεται. 22 Φεβρουαρίου θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και ο καθένας θα προσπαθήσει στα πλαίσια αυτά να έρθει σε συμβασμούς κλπ. Τελειώσαμε με το σημείο αυτό της ημεσίας διάταξης. Πάμε στο τελευταίο μας σημείο για σήμερα το απόγευμα. Η κυρία Λίν θα λάβει το λόγο για να μας παρουσιάσει γρήγορα, μα πάρα πολύ γρήγορα, μια πρόταση ψηφίσματος που έχει να κάνει με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομιακό και υγειονομικό τομέα. Ο Δήμος Ροπ ε, διαμαρτυρήθηκε ο εκπρόσωπο ότι μεταξύ των κοινωνικών τρόπων δεν τηρούνται συμφωνίες, Νομίζω ότι πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση και δίνουμε το λόγο και στη διαδικασία αυτή όμως δεν δεχτήκαμε μόνο μια προφορική, μόνο προφορικές τροπολογίες γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε αύριο στο σχέδιο ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Ξέρουμε ότι περίπου ένα εκατομμύριο είναι οι τραυματισμοί από βελόνες ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι εργαζόμενοι στον τομέα εργασίας περιμένουν μήνες και μήνες με αγωνία μεγάλη για να δούνε αν έχουν υποστεί λίμωξη ή όχι μετά από τον τραυματισμό. Έχουμε δουλέψει ε, επανειλημμένα πάνω η ώρα να οδηγηθούμε σε κάποιο συμπέρασμα. Το 2006 ε, είχαμε μία οδηγία και ο Στίβεν και εγώ είχαμε υποβάλει ε, τότε με συγκεκριμένες τροπολογίες Υπάρχει και άλλο ψήφισμα του 2008 βάσει της ε, οδηγίας ε, για την έκθεση σε βιολογικούς ε, παράγοντες και για εργαζόμενους που διατέχουν κίνδυνο λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες. Όμως περιμένουμε τελικά μέχρι να υπάρξει πρόταση της Επιτροπής έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους πιστεύουμε ότι αργήσαμε πολύ και πιστεύω ότι έστω και αν πραγματικά νομίζω ότι οι συμφωνίε με τους κοινωνικούς εταίρους είναι κάτι σημαντικό, ε, παρόλα αυτά πρέπει να κινούμαστε και γρήγορα. Ε, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους της τις τροπολογίες. Είχα τροπολογίες από το ΕΛΚΑ, από τους σοσιαλιστές ε, και από το, τους Ευρωπαίους Δημοκράτες και μεταρρυθμιστές εκτός από μια αλλαγή η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί, δηλαδή να μην γίνει αναφορά ε, στο άρθρο 1α του FTAU ε, στο, ε, στην τροπολογία 4, γιατί όντως είναι το τομεακό και συμφωνήσαμε ότι συνήθως δεν αναφέρουμε τέτοιου είδους πράγματα, άρα δεν υπάρχει λόγος και εδώ. Δεν ξέρω εάν κάποιο θέλει να πάρει το λόγο, πάντω εγώ αυτά ήθελα να πω. Δεν euh, ξέρω αν επιθυμούν τα μέλη. Δύο μέλη είναι για γραμμένα. Να σας ευχαριστήσω γιατί δείξατε στη συζήτηση αυτή με τους κοινωνικού εταίρους τι ακριβώς γίνεται. Εδώ καμιά φορά όταν είμαστε πιεσμένοι τα πετυχαίνουμε όλα αυτά και Ίσως μερικές φορές να επιτυχεί με την διαδικασία, αλλά οι δύο προσεγγίσεις είναι συμπληρωματικές και απαραίτητες, διότι μία δεν επαρκεί και δεν αντικαθιστά την άλλη. Σαρκάς και Μπαλντασάρ. Σύντομα, σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει την κυρία Λίνα να την συγχαρούμε για αυτό το έγγραφο και έτσι μπαίνουμε στα πλαίσια αυτής της συζήτησης, έστω τώρα στο τέλος αλλά ακριβώ αποδίδει δικαιοσύνη στην εργασία μας του Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή που έτσι μας επέτρεψε να εκφράσουμε την απόψή μας και τον κύριο Χιούς που εργάστηκε πολύ γι' αυτό, να τον υπενθυμίσουμε λοιπόν και ε, θα πρέπει να τα πούμε αυτά πράγματα σε μια παρόμοια στιγμή. Όπως σήμερα το Κοινοβούλιο βοηθάει ακριβώς τους κοινωνικούς εταίρους και αναγνωρίζει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όλα αυτά που κάνουμε όλοι μας μαζί ελπίζω να αποτελούν επιπλέον στοιχείο ώστε να ανταποκριθούμε στα όσα απαιτούν από εμά με ένα κοινωνικό πρότυπο ευρωπαϊκό που να είναι αναγνωρίσιμο από τον μέσο πολίτη. Κύριος Μπαλταζάρ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ σύντομος σύντομο θα είμαι, σαν σκιώδη συγητής από ΕΛΚ. Να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την πρόταση αυτή ψηφίσματος. Νομίζουμε ότι το θέμα που θίγει είναι πολύ ευαίσθητο και είναι κάτι το κατεπήγον αυτό για τους εργαζόμενους στη, παρόλο στον τομέα αυτό με ένα εκατομμύριο τουλάχιστον άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε ικανοποιημένοι που επιμένουν επιτέλους δεν κάνει κάτι η Επιτροπή αλλά οι κοινωνικοί εταίροι πέτυχαν μια συμφωνία και νομίζω ότι αποτελεί τον σωστό τρόπο αυτό έτσι για να προχωρήσουμε και ε, και να συνεχίσουμε και με παρόμοια ψηφίσματα για να υπάρξουν οι αποφάσεις. Αποτελεί λοιπόν προηγούμενο σωστό και καλό. Έχουμε τι μαζί με τις συνεισυγήτρια δεν είχαν να κάνουν με τον κεντρικό πυρήνα του ψηφίσματος, απλά και μόνο ισχυροποιούσαν ορισμένες απόψεις. Πάνω απ' όλα το ελάχιστο αυτό που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία επιτρέπει στα κράτη-μέλη από τη στιγμή που το επιθυμούν να υιοθετήσουν και αποφάσεις mm. θετικότερες και ψυχολότερου περιεχομένου. Το επιθυμούμε αυτό και ταυτόχρονα όμως τώρα δεν θα έπρεπε να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα το ψήφισμα αυτό. Μπορούμε να εκφράσουμε λοιπόν μια κάποια ικανοποίηση για την εργασία. Την ικανοποίησή μας ε, για την εργασία αυτή και να σας πω ότι χρειάστηκε να θίξουμε αυτό το σημείο στο κείμενο ότι θέλουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη αυτής της συμφωνίας. Πολύ συχνά εμείς ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό και επιθυμούμε λοιπόν να έχουμε συνεχή ενημέρωση. Η κυρία Φιγκερέιντο και μάλιστα σύντομα σύντομα σας παρακαλώ. Πρόεδρε σας ευχαριστώ. Σύντομα πραγματικά να πω κάτι γιατί και εμείς θα θέλαμε να υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή. Νομίζουμε ότι θίγει τα βασικά σημεία. Βέβαια, πάντα μπορεί κάτι να βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν ε, τα κύρια σημεία και η συνάδελφος Λίν έκανε πολύ καλή εργασία ό,τι γινόταν στον τομέα αυτό τώρα. Ευχαριστώ. Κανονικά είχε κλείσει ο κατάλογος στον μιλητό, αλλά εδώ ο συνάδελφος ζητάει το λόγο. Σύντομα, σύντομα έχει το λόγο συνάδελφε. Σύντομα, σύντομα. Να πω ότι συμφωνούμε με αυτή τη συμφωνία και εμείς δεν υπάρχει καμία επιφύλεξη για την γνωμότητα της κυρίας Λίν και εντάξει μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Αλλά λοιπόν βλέπω ότι συμφωνούμε, δεν χρειαζόμαστε τις διευκρινήσεις της Επιτροπής. Να, μια φορά που συμβαίνει αυτό, αλλά η συγγήτρια έχει το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Απλώς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία. Κρίμα που ο Στίβεν Χιούς δεν μπόρεσε να είναι παρόν, γιατί εμείς οι δυο δουλέψαμε επί χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα. Ελπίζω το Συμβούλιο τώρα, από τη στιγμή που το περάσουμε εμείς, θα προωθήσει το θέμα αυτό και δεν θα υπάρχουν πλέον τραυματισμοί από αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία μπορούμε να, τα να τους προλάβουμε τους τραυματισμούς. Ευχαριστώ. Αύριο το πρωί θα το πούμε